Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες σήμερα, σειρά ψηφοφοριών. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας για να ψηφίσετε. Και η Λίντα Μακάβαν. Θέλει να πει τίποτα. Thank you, thank you, Chairman. We've arrived this morning. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φτάνοντας εδώ, ανακαλύψαμε κάτι χαρτιά από λόμπι, κάτι που λέγεται συμμαχία για τη διαφάνεια και κάτι τέτοια. Όλοι ξέρουμε τις ομάδες πίεσης εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν νομίζω πως είναι αποδεκτό να βρίσκουμε εδώ έγγραφα από τα διάφορα λόμπι εντός των ενθούσεων. Ζητώ λοιπόν από τη Γραμματεία να μην επιτρέπουν στους διάφορους εκπρόσωπους των ομάδων πίεσης να έρχονται εδώ και να μας μοιράζουν χαρτιά. Καλύτερα να τα στέλνουν στα γραφεία μας, άμα θέλουν να μας στείλουν πληροφορίες. Yeah, that's... Συμφωνώ. Την επόμενη φορά να προσέχουμε, η γραμματεία δεν είδε τίποτα. Από ό,τι φαίνεται μπήκανε πριν έρθει κανείς. Η Ντάκμαρ για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στο ίδιο πράγμα. Είμαστε αυτήν την Επιτροπή εδώ και πάρα πολύ καιρό και φυσικά έχω επαφέ με διάφορε ομάδε ε, συμφερόντων ε, από εξαπανέκαθεν αλλά ε, και βρίσκω ότι οι ευρωβουλευτέ ε, πάντοτε έχουν επαφέ με τι ομάδε πίστη και είναι και φυσιολογικό. Όμω εδώ γίνονται διάφορε απόπειρε πολύ άσχημε, Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα νέο κώδικα δεντολογίας για να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε με τις επαφές μας με τον εξωτερικό κόσμο και τι επαφέ μα με τι ομάδε πίεσης. Εγώ πάντοτε ήμουν πολύ ήπια, λέγοντας ότι το χρειαζόμαστε την επαφή με τις ομάδες πίεση. Αλλά από εδώ και μπρο, οποιοδήποτε συμπεριφέρεται έτσι, ε, ε, επιβαρύνει ολόκληρο τον κλάδο των ομάδων πίεσης, γιατί είμαι βέβαιη ότι το Προεδρείο τώρα θα φτιάξει πολύ αυστηρού κανόνες πρόσβασης. Οποιοδήποτε σκέφτηκε λοιπόν πω ήταν καλή η ιδέα αυτή, ε, θα το μετανιώσει. Καλώς. Εγώ διαμαρτύρομαι. Εμένα δεν μου δώσαν τίποτα στο Προεδρείο. Δεν είχαν προβλέψει χαρτιά για το Προεδρείο. Εν πάση περιπτώσει, λήφθη το μήνυμα και ε, θα προσέχουμε την άλλη φορά. Σας λέω, ήρθανε πριν μπει κανείς στην αίθουσα πολύ νωρίς. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Περιορισμό χρησιμοποίηση ε, ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικέ και ηλεκτρονικέ συσκευέ. Αναδιατύπωση λέει εδώ. Η Σάτου Χάση ζήτησε το λόγο προσωπώντα την συγκεκριά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Εύανς που είναι η συγκήτρια και η οποία δεν μπορεί να παρευρεθεί προς το παρόν. Το θέμα εδώ είναι το εξής. Μάλλον το, η αναδιατύπωση γίνεται, η διόρθωση αυτή γίνεται με σκοπό να ευθυγραμμιστούν οι ε, διατάξεις αυτές στο νέο κανονισμό των ε, εφαρμοστικών πράξεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει την θέση του σε πρώτη ανάγνωση πριν τεθεί σε ισχύ αυτός ο κανονισμός ε, την 1η Μαρτίου. Όμως η δημοσίευση της οδηγίας δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί μέχρι τότε. Γι' αυτό η νομική υπηρεσία και των του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου θεωρούν ότι οποιαδήποτε πράξη που έχει δημοσιευθεί μετά την ημερομηνία αυτή, μετά την 1η Μαρτίου του 2011, δεν μπορεί να θεσπίζει διαδικασίες με βάση την προηγούμενη απόφαση επιτροπολογίας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να προσαρμοστούν ανάλογα ε, αυτές οι διατάξεις, γι' αυτό ζητείται η διόρθωση ή διατύπωση. Äh, Ευχαριστώ. Μία ψηφοφορία λοιπόν. αμέσω αρχίζει τώρα ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Υπερκατά δεν λέω. Abstimmung ist 56. Κανείς κατά καμία αποχή ομόφωνα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία εισηγήτρια. Και συνεχίζουμε το σημείο 9. Και αυτό είναι διόρθωση για τα πλαστά φάρμακα ή παραποιημένα όπως λέω. Μία ψηφοφορία μόνο, ηλεκτρονική. Αρχίζει τώρα. Abstimmung Πέρας ε, της ψηφοφορίας. Ομόφωνα. 54 υπέρ, κανείς ε, κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Συνεχίζουμε. Είναι λίγο μεγαλύτερη αυτή η ψηφοφορία τώρα. Τροποποίηση οδηγίας που αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην επικράτειά τους. Η Κορίν Λεπάζη, συγγήτρια. Και έχουμε πρώτη που ζήτησε το λόγο την κυρία Κορτίνες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προειδοποιήσω. άλλη συνάδελφος ε, είχε αυτό το θέμα, η οποία έχει αποχωρήσει, δεν είναι πια βουλευτή ε, και την ευχαριστώ για τη δουλειά τη, αλλά πρέπει να σα πω ότι δεν είχαμε χρόνο να το επεξεργαστούμε στην ομάδα όπω έπρεπε. Ε, ήθελα και ζήτησα επανειλημμένα να αλλάξει η ημερομηνία ψηφοφορία για να έχουμε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε. Για ποιο λόγο, Γιατί πιστεύω ότι θα έπρεπε να βελτιωθεί το κείμενο για να μην έχει προβλήματα στο Συμβούλιο. Τώρα θα βρούμε το Συμβούλιο μπροστά μα. Έχει πάρα πολλέ επαναλήψει. Ε, πάρα πολλές βελτιώσεις χωράνε. Και η ομάδα μου αισθάνεται πάρα πολύ άβολα ε, γιατί άρον-άρον θα πρέπει να ψηφίσουμε το σημαντικό έγγραφο χωρίς να το έχουμε επεξεργαστεί όσο θα οφείλαμε. Ευχαριστώ. Η συγκήτρια, παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι θα ε, ψηφίσουμε επ' αυτού του κειμένου, το οποίο αποτελεί πρόταση της ε, Επιτροπής με στόχο να δοθεί περισσότερη ελευθερία στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να περιορίζουν τη φύτευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω θερμότατα ολόκληρη την ομάδα της διοίκησης, τους συνεργάτες μου και κυρίως τον Σκιώδη Συγητή. Συνεργαστήκαμε επανειλημμένως για να ολοκληρωθεί το κείμενο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκουτιέρες, η οποία καθοδόν ενεπλάκη στην προετοιμασία. Δεν ήταν πολύ εύκολο για αυτήν. Είπε ότι θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Θα μας άρεσε να αναβληθεί ε, για οκτώ ημέρες η ψήφιση αυτού του κοινοβουλίου, του κειμένου, για να μπορέσει ε, να μελετήσει το ΕΛΚ. Δεν μπορέσαμε να το βάλουμε στο 18 γιατί υπάρχει το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών και θα έμπαινε στο τέλος του μήνα και θα τροποποιούσε τελείως την ημερήσια διάταξη. Ήταν πάρα πολύ μακριά. Γι' αυτό διατηρήθηκε η ψηφοφορία σήμερα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τέλειο, αλλά ποιος είναι τέλειος. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στο, εδώ ενώπιόν μας ένα σχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ισόρροπο. Λαμβάνει υπόψη του τις διάφορες ε, ε, απόψεις που πολλές φορές δεν είναι εύκολο να γίνει. Πρόκειται για ένα κείμενο που χορηγεί περισσότερη ελευθερία στα κράτη-μέλη. Μας ενδιαφέρει όμως επίσης να υπάρχει ένα κοινοτικό κατόφλι, ε, μια κοινοτική αξιολόγηση. Και πιστεύω ότι με αυτό το κείμενο αυτό επιτυγχάνεται. Δεύτερον, υπάρχει με αυτόν τον τρόπο περισσότερη νομική ασφάλεια. Γι' αυτό τροποποιήθηκε η νομική βάση και ταυτόχρονα σκοπός μας ήταν να μην φυγούν οι κανόνες της εσωτερική αγοράς. Κατά τρίτον, φροντίζουμε να τα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2008, τα οποία είμαστε προσιλωμένοι, να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Αυτό έχετε ενώπιόν σας. Είμαι ιδιαίτερος ε, ευγνώμων για όλους όσοι ασχολήθηκαν επί ώρες για να βρεθούν αυτές οι συμβαστικές λύσεις τις οποίες τελικά καταλήξαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λοιπόν, έχουμε τρεις τροπολογίες που μάλλον ταυτίζονται οι τρεις πρώτες. Η Σαμπίνε Βέλης έχει αποσύρει το όνομά της από τη 12, το έχει κοινοποιήσει. Λοιπόν, ψηφίζουμε τις τρεις μαζί. Ψήφι κατά αποχές απορρίπτονται. Ακολουθεί Α, τι είναι αυτό που λέει εδώ, συμβιβαστική, ένα, ψήφι Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα είναι μια άλλη consolidated, δηλαδή δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη παρακαλώ 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική παριθμό 4 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική παριθμόν 6 κατά αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημένη, όχι συμβαστική. Ενοποιημένη 7 ψήφι π. Κατά αποχές εγκρίνεται επίση. Η ενοποιημένη 8 ψήφι π. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ, καλά, να το ελέγξουμε τότε. έφνετ. Άρχεται η ψηφοφορία για την οκτώ ενοποιημένη. Also ein PPE zu viel, ein SO... Περσεύει ένα ΣΕΛΚ και ένα σοσιαλιστή. Ein S&D zu viel και σοσιαλιστής και δημοκράτης. Πέρας. 31 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. Τι έγινε, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω την κάρτα ψηφοφορίας. Μπορείτε να καταγράψετε την ψήφο μου. Μα όταν κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτό που ισχύει είναι ότι ψηφίζετε ηλεκτρονικά και λυπάμαι. Στείλτε να σας φέρουν. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Βοηθούς δεν έχετε. Σε πέντε λεπτά η βοηθός σας έχει επιστρέψει με την κάρτα ή ο βοηθός. Αξίζει τον κόπο. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Λοιπόν, ε, συμβιβαστική υπαριθμών 9. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται ή ενοποιημένη υπαριθμών 10 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημένη 11 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές πε. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημενη 11 ψηφι πε, κατα αποχες εγκρινεται ενοποιημενη 12 υπερ κατα αποχες εγκρινεται η συμβιβαστικη 13 ψήφι πε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική, συγγνώμη, ενωπημένη 14 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ενωπημένη 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημένη 17 υπέρ. κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε το διατακτικό. Τα άρθρα δηλαδή. Ε, 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 56 υπέρ. Α, τσεκ θέλετε για την 55, τι λέξουμε. Το ΕΛΚ είναι πολύ πρόθυμο και θουσιώδες, αλλά έχει τρεις βουλευτές παραπάνω. Τώρα εντάξει. Πέρασε. Είναι Εγκρίνεται. Η 56 Ψηφί υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια. δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στη σελίδα 6 λέει τώρα. Ε, Άγκρι 9. Μισό λεπτό να το. Στην 84. Σελίδα 6. Κάτω-κάτω είναι η τροπολογία 84. Ψήφι Κατά αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ερχόμαστε στη σελίδα στιγμή να τη βρω. Κερδίσαμε πολύ με τις συμβιβαστικέ. Seite 14. Σελίδα 14 είμαστε τώρα. Ταυτίζονται 86, 87 και η 12 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ των τριών αυτών. Κατά. Α, χρειάζεται παλήθευση αυτό. Λοιπόν, ας το επαληθεύσουμε. Πέρας. Ναι, ήταν μικρή διαφορά, απορρίπτεται, 29-31. Γυρνάμε σελίδα. 88, ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. Seite 17. Στη σελίδα 17, 99 και η 13 της Γεωργίας είναι ταυτόσιμες. Ο Πίτερ Λίζε, μια παράκληση. Δεν έχουν όλες οι πολιτικές ομάδες τις ίδιες σελίδες στον κατάλογο ψηφοφορίας. Μπορείτε να μην μας λέτε σελίδες, αλλά αριθμό τροπολογίας. Ωραία, ευχαριστώ για τη συμβουλή. Σε μένα είναι σελίδα 17. Τώρα στη δικιά σας λίστα δεν ξέρω πού τη δέχετε. 99 και 13 ε, της Γεωργίας. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πάμε στην τροπολογία Μπερθμον 100, έτσι δεν είναι. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. Η 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Γιατί είναι 103 παρακαλώ. beendet. Πέρασε. Απορρίπτεται. Λείπει η κάρτα της συναδέλφου Μάνερ, αλλά τι να κάνουμε, δεν αλλάζει αυτό τώρα, τελείωσε. Η 14 της Επιτροπής Γεωργίας. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Ωραία, στο ελέγξουμε. Τη 14 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά της Επιτροπής Γεωργίας. Περσεύει ένα σέλκ ακόμα. Βγάλτε μία κάρτα από το Λαϊκό Κόμμα σας παρακαλώ. Τώρα είμαστε εντάξει. ist vorher. angenommen. Also. Εγκρίνεται. Ναι, αλλά δεν σηκώνατε χέρια. Πού να το καταλάβω. 108 και 109 ταυτίζονται ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ χρειάζεται παλήθευση νομίζω. Ε Το ΕΛΚ έχει ακόμα μία κάρτα παραπάνω. Εντάξει. Απορρίπτεται με ισοψηφία παρακαλώ. 110. Ρενάτη Σόμερ. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 της Γεωργίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Η 17... όχι, 112 ψήφι υπέρ. Η 7 τη Γεωργία κατέπεσε. Ε, κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά Αποχέ απορρίπτεται. 114 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 της Γεωργίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ Dagegen. κατά αποχές εγκρίνεται. Οι αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Ε, τροπολογία 13, υπέρ. Κατά. Άποχες, έλεγχος. Για τη 13, παρακαλώ, απελευθεύουμε ηλεκτρονικά. Und beendet. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Και πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 22. Αιτιολογική σκέψη 2α νέα. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας 22. Κατά. Αποχές. Έλεγχος χρειάζεται και εδώ. Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελειώνει. Απερίφθη. 23. Ψήφι υπέρ. Υπέρ της 23. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και συνεχίζουμε αιτιολογική σκέψη 9α, η τροπολογία 53 του κυρίου Παλέτσκης. Ε, ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίφθεται. Η 54 του ιδίου είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάσαμε ήδη στην τελική ψηφοφορία. Μα είναι θαυμάσια όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Ηλεκτρονικά λοιπόν ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Ακόμα περισσεύει ένα σελφ. Abstimmung beendet. Πέρας. 34 υπέρ, 9 κατά, 17 αποχές. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ, 10 ε, κατά, 16 αποχές. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για όλη τη δουλειά της και βλέπουμε ότι χρειάζεται κάποια συζήτηση ακόμα για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάντως ήταν μεγάλο το θέμα και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη γραμματεία μας.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 So, dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Änderungs, also Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ψηφοφορία που είναι το σημείο 11 στην ημερησία διάταξη κοινή γεωργική πολιτική με χρονικό ορίζοντα το 2020. Διατροφή, φυσική πόρη, έδαφος, μελλοντικές προοπτικές και προκλήσεις. Η συγκήτρια είναι η κυρία Κάντενμπαχ. Έχουμε μερικές αλλαγές τις οποίες και θα σας ε, αναφέρω όταν θα φτάνουμε εκεί. Αρχίζουμε. Τροπολογία παριθμών 11. Κρίστα Κλάς και ε, ε, λυπή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Zufrieden δεν είστε ικανοποιημένοι. Ο κύριος Σνέρχαρτ θέλησε να με διορθώσει. Αλλά είναι πολύ χαρούμενος που εγκρίθηκε. Να πέσει. Ε, τι θέλει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τη συμβιβαστική υπαριθμόν 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 7. Έχουμε χωριστή ψηφοφόρια. Το πρώτο τμήμα ψήφιπε Κατά τμήματα καλύτερα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το άλλο τμήμα ψήφι Κατά. Αποχές έλεγχος. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 7. Τι θα γίνει με το ΑΕΛΚ, ακόμα δεν περισσεύει ένας. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 9. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 12. Υπέρ. Κατά. Χρειάζεται παλήθευση εδώ, δεν βλέπω καλά. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Dagegen Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 2 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημένη τρία τώρα, ψήφιπε. Κατά. Α, ναι, σωστά. Δεν το είχα δει. Είναι χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα. Τμήμα πρώτο, είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για το δεύτερο λοιπόν τμήμα αποζητάτε. Για τους απίστους. Το ΕΛΚ συνεχίζει ένας παραπάνω. Πέρας. Εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. Στη 30, στον Καστόν Φραγκό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες πώς ψήφισαν υπέρ, κατά, δεν είδα. Α, αν είναι υπέρ, εγκρίνονται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η ενοποιημένη 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Η 56. Ελένα Ωνα Αντωνέσκου, υπέρ. Παρακαλώ. Ισά του χάσει. Η ομάδα μας θεωρεί η τροπολογία μας 51 και αυτή θα πρέπει να εγκριθεί γιατί η συμβιβαστική τροπολογία 3 δεν καλύπτει ούτε αυτήν ούτε την τροπολογία 45. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει γίνει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοριών σε σχέση με αυτές τις δύο ψηφοφορίες. Λοιπόν, επειδή το δεύτερο τμήμα της ενοποιημένης τροπολογίας 3 εγκρίθηκε, φρονούμε ότι η 51 καταπίπτει. Το ίδιο δεν ισχύει και για την 45. Συνεχίζουμε. Στην 56 ήμασταν της κυρίας Αντωνέσκου, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Η 39 Μακάβαν ψηφίπε. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 40. Ορέστε Ρώση υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Γιατί 40. Πέρας. Γκρίθηκε. 41 είπε Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 43 είπε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 47. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, ήταν χωριστή η ψηφοφορία, άρα τι ψηφίσαμε τώρα, το πρώτο τμήμα μόνο. Oh no, sorry, sorry, sorry. Nee, es geht mit 55 weiter. Also, Änderungsantrag. 55 τώρα. Χωριστή ψηφοφορία, τμήμα πρώτον. Ψηφιπέ. Κατά. Άποχες, απορρίπτεται. Το δεύτερο, υπέρ. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Μάλιστα. Οπότε ψηφίζουμε τη C6 ενοποιημένη. Η κυρία Κάντεμπαχ αποσύρει την υποστήριξή της, παρόλα αυτά θα την ψηφίσουμε. Ε, ψήφι υπέρ της ενοποιημένης 6. Κατά. Αποχές, έλεγχος. Αρχίζει ψηφοφορία. Δύο παραπάνω στο έλκτο. τώρα. εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται η ενοποιημένη έξι. Και ψηφίζουμε με μονομένα τις τροπολογίες. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος για την 57. Πέρα. Εγκρίνεται. Η 59, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 63 χωριστή ψηφοφορία, τμήμα πρώτο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 64-65 υπέρ και τις δύο μαζί τις ψηφίζουμε γιατί είναι ταυτόσιμες. Κατά αποχές εγκρίνονται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 73 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Η 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 77, 78, 79, 80, 81 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 82 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Αφού εγκρίθηκαν οι προηγούμενες, μάλιστα. 84 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 86 σε τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, συγγνώμη, 87 διορθώνει ο πρόεδρος, 87 του κύριου Αρσένη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ή 88 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8, όχι πώς τη λένε την άλλη, ενοποιημένη 8 υπέρ. Α, και σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον. Ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συνεχίζουμε. 93 ε, ναι, τώρα. Ψήφιπε. Κατά. Απόχες. Νομίζω ότι έχει ελεγχθεί, αλλά, ε, εγκριθεί, αλλά χρειάζεται έλεγχο, παρακαλώ, για την 93. Πέρασε. Ναι, εγκρίνεται. 94. ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Υπέρ. Σε 99. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτη 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 101 είπε. Η ΣΑ του χάσει ζητάει το λόγο για την 101. Έχω μια προφορική τροπολογία για αυτή και για την επόμενη τροπολογία. Διαβάζω την τροποποιημένη εκδοχή της τροπολογίας ανησυχεί για την οικολογική κατάσταση ευρωπαϊκών υδάτινων μαζών, στις οποίες καταλήγουν τα ύδατα από γεωργικές περιοχές, όποτε, όποτε είναι προφανές ότι δεν τηρούνται βασικά κριτήρια εφορίας. Για παράδειγμα, στη Βαλτική θάλασσα, που είναι μία από τις πλέον μολυσμένες θάλασσες του κόσμου, επισημαίνει ότι η γεωργία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές ισρών, μεγαλυτερες πηγες εισρων αντι τη μεγαλύτερη πηγή θρεπτικών ουσιών κτλ. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσω και την προφορική τροπολογία της επόμενης, του επομένου κειμένου, της τροπολογίας 102. Ζητάμε να διαγραφεί ο όρος κλειδί πριν από α, τους βασικούς στόχους. Αντί key objectives, βασικούς στόχους, να λέει σχέ, απλώς στόχους. Μάλιστα, πρέπει να ρωτήσω. Διαφωνεί κανείς να εγκριθεί η προφορική τροπολογία για την 101. Διαφωνεί κανείς να δεχτούμε αυτή την προφορική τροπολογία. Για την 102 ποιος διαφωνεί με την προφορική τροπολογία μπορούμε να την ψηφίσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία της Άτου Χάση ψήφι υπέρ όχι την προφορική γιατί υπήρξε αντίρρηση. Κατά αποχές απορρίπτεται. 102. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε χωρίς το βασικές υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 104 κατά τμήματα. Τμήμα πρώτο είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 είπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και ερχόμαστε τώρα στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει. Πέρας. 59 υπέρ, ομόφωνα, χωρίς αποχές και αντίθετες ψήφους. Ε, συγχαρητήρια, Κάριν Κάντεμπαχ ομοψυχία της Επιτροπής Περιβάλλοντος που από κοινού θα επερασπίσουμε στην Επιτροπή Γεωργία στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερα δεν γίνεται από ομόφωνα, πόσο καλύτερα να γίνει. Και ερχόμαστε στο σημείο 12 τώρα. Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων Πάβελ ποτ είναι ο εισηγητή και ψηφίζουμε. Έχουμε τι 41, 42 και 43 τροπολογίες που ταυτίζονται, ψήφι υπέρ και των τριών. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 44 υπέρ. Κατά αποχές Σαν 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 επερ. κατα κατά αποχές εγκρίνεται 51-52 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 53 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 1 είναι γλωσσική και ερχόμαστε στην 61 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Άποχες. Πράσινα χέρια δεν είδα. Ελέγχουμε την 64. Πέρασε. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Άποχες εγκρίνεται. 68 Έχει προφορική τροπολογία εδώ. Υπέρ της 68 με την τροφο... προ... προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 68 παρακαλώ να ελεγχθεί ηλεκτρονικά. Ακόμα περσεβαίνεις από το ΕΛΚ. Ψηφίζει ένας παραπάνω στο ΕΛΚ από όσους δικαιούνται. Τώρα εντάξει. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Και ψηφίζουμε το κείμενο χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ, την αρχική 68 δηλαδή, κατά αποχές. Και πάλι χρειάζεται παλήθευση αυτό, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν άλλαξε τίποτα και πάλι στο ψηφίο και απορρίφθηκε. 69. υπέρ. Κατά. Αποχές, γκρίνεται. 70, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 71 υπέρ. Κατά. Αποχές, απο, ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 73 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Οι άντρες φιλελεύθεροι δεν σηκώνουν χέρι. 74. Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 Είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 Είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 79 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 80 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 81 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 82 επέ. Κατά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 αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101. Α, για την 100 θέλετε έλεγχο. Καλώς. Πέρας. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ Κατά. Yeah. Α, έχει καταπέσει εφόσον εγκρίθηκε η προηγούμενη. Λοιπόν, απερίφθη όμως η 103, οπότε γι' αυτό ψηφίζουμε την 105. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 105. Σύρπα τι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Καλά. Πέρας. Έχει απορριφθεί. Φία. Για 104 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 καταπίπτει και πάμε στην 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Dagegen. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116, 117. 116, 117. Κατά. 118, η προηγούμενη απερίφθη. 18 υπέρ, 118. Κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Στις αιτιολογικές σκέψεις ερχόμαστε τώρα. Η τροπολογία 7, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 15 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος. Γιατί 19. Abstimmung Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Τι θέλετε, έλεγχο για την 36, καλώς. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 36 αρχίζει τώρα. Και τελειώνει επίσης. Εγκρίνεται. 38 είμαστε τώρα, έτσι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, Ας ελέγξουμε την 6 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε. Απερίφθη μάλιστα. Ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική αρχίζει τώρα. So, 12 κατά, 29 υπέρ, 17 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά και ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Στην μέση διάταξη. Ο κύριος Σόμερ που είναι. Ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Έχει αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία όμως για την άλλη εβδομάδα. Αλλά μας δίνει αυτό την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε αυτό το περίπλοκο θέμα. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα το πρωί την ώρα που έχουμε την ευκαιρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, δίνω το λόγο στην κυρία Στρόμαρ που είναι η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήταν χρήσιμο και ευγενικό αν κάθονταν οι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σερ κολέγκα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφοφορία της έκθεσης μου για τη σήμανση των τροφίμων, όπως γνωρίζετε, αναβλήθηκε για την άλλη εβδομάδα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η αρχική ε, ημερομηνία ε, ήταν αυτή. Προσπαθήσαμε να την προτάξουμε για τούτη τη εβδομάδα, αλλά αυτό δυσκόλυψε πάρα πολύ τη γραμματεία και εμάς κατά τα άλλα, πρέπει να σας πω, διότι ε, οι μεταφράσεις έφταναν πάρα πολύ ε, διστακτικά και αργά. 400 τροπολογίες παρακαλώ έχουν κατατεθεί και οι τελευταίες ε, μεταφράσεις από ό,τι γνωρίζω έφτασαν εχθές το βράδυ. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί το θέμα του παραδεκτού βέβαια των τροπολογιών. Ε, δεν έχει τελειώσει αυτό Οι κανόνε είναι σαφείς, σαφέστατοι ε, για τη δεύτερη ανάγνωση, τι είναι παραδεκτό και τι όχι. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται βουλευτές που δεν είναι μέλη της ε, αρμόδιας επιτροπής να κάνουν τροπολογίες, γιατί είχαμε και τέτοια περιστατικά. Επίσης δεν μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες για θέματα που απερίφθησαν στην πρώτη ανάγνωση αλλά για το κατά πόσο είναι παραδεκτές ε, ε, όλες οι τροπολογίες δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Από την περασμένη συζήτηση ε, κοιτάξαμε τα βασικά προβλήματα που έχουμε για τη δεύτερη ανάγνωση. Θα τα ξαναπώ και σήμερα γιατί είναι περισσότεροι παρόντες συνάδελφοι από ό,τι την περασμένη φορά. Το πρώτο πρόβλημα είναι η σήμανση στην πρόστια πλευρά της συσκευασία και το δεύτερο η ε, σήμανση της προέλευσης των τροφίμων. Mm-hmm. Στην πρόστια όψη λοιπόν έχει ως εξής η κατάσταση. Στην πρώτη ανάγνωση αποφασίσαμε να αναφέρεται και η ενεργειακή αξία, οι θερμίδες δηλαδή, και οι θρεπτικές ουσίες, τα συστατικά του προϊόντος ε, για τα άλατα, για τα σάκχαρα, για τα κορεσμένα λίπη. Το Συμβούλιο κάθετα το απορρίπτει αυτό. Και σου λέει ποια είναι η προστινή πλευρά του τροφίμου, γιατί υπάρχουν τρόφιμα που από τη συσκευασία τους ε, έχουν πολλές πλευρές τις οποίες θα μπορούσε κανείς να εκλάβει ως πρόσθεια πλευρά. Ε, ε, και πρότεινα ένα ορισμό εγώ. για να αναφέρει την ενεργειακή αξία και άλλοι συνάδελφοι έχουν φέρει και άλλες τροπολογίες μετά την πρώτη ανάγνωση για επιπλέον θρεπτικά συστατικά κτλ. Μπορώ να φανταστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτό το καιρό γίνεται ένα τεράστιο λόμπι για να αναφέρονται οι μερίδες. Τεράστια πίεση. Με τέτοια επιθετικότητα δεν έχω ξαναζήσει εγώ τέτοιο λόμπι και το θεωρώ και ανάρμοστο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους συναδέλφους, γιατί ξέρω ότι τους πιέζουν και εκείνους. Ε, αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται πια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναγράφεται επιπλέον η, η μερίδα, στην προστινή πλευρά. Ε, μαζί με την ενεργειακή αξία, αλλά ανά 100 γραμμάρια ή ε, μιλιλίτρε προαιρετικά. Δεν αποκλείω τίποτα. Αυτό το θέμα όμως της, θερμή, της μερίδας ποιο είναι. Ακριβώς το ίδιο όπως και στο παρελθόν. Το μέγεθος της μερίδας δεν ορίζεται. Οπότε ε, μπορούν οι παραγωγοί και οι κατασκευαστές να επινοούν μία μερίδα ε, για προϊόντα που έχουν πολλές θερμίδες και πολύ ενεργειακή ε, μεγάλη αξία για να φαίνεται στη μερίδα ότι έχει λίγες θερμίδες. βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα που λέει να βάζουν και πόσο είναι η μερίδα εθελοντικά. Ναι, αλλά αυτά συνήθως τα βάζουν στην πίσω πλευρά της συσκευασία. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η σήμανση προέλευσης των προϊόντων. Εκεί ε, κατατέθησαν πάρα πολλές τροπολογίες και είναι ένα χάος και το προσπαθώ να βάλω λίγη τάξη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές τομεακές κλαδικές ρυθμίσεις για τη σήμανση της προέλευσης των τροφίμων, για φρέσκα φρούτα και λαχανικά παράδειγμα, ή και για τα ψάρια. Επίσης στο γάλα θα ήταν καλύτερη μια ε, τομεακή προσέγγιση, πια μια εγκάρσια τελεία, ε, ε, τελείω συγγνώμη, στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Συστηματικά είναι καλύτερο να έχουμε ανακλάδο προσέγγιση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να προτείνει το Συμβούλιο υποχρεωτική σήμανση, υποχρεωτική και για πρόβατα, χείρους και πουλερικά, το κρέας πάντα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κάτι ακόμα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι παρεξήγηση. Το διαπίστωσα σε πολλές συνομιλίες που είχα και βέβαια θα υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ε, για όλα τα προϊόντα που μπορεί κανείς να φανταστεί, έθελοντικά να δηλώνει ε, κανείς ε, προέλευση, ακόμα και την περιφέρεια. Να μην είναι όμως παραπλανητικό για τον καταναλωτή. Δηλαδή εθελοντικά να μπαίνει μια ετικέτα που να παραπλανεί τον καταναλωτή και να νομίζει αυτός ότι έρχεται από κάπου αλλού το προϊόν και όχι από εκεί που είναι. Εθελούσε είναι όλο αυτό. Επίσης και στα κατεργασμένα προϊόντα ε, να αναφέρεται το κύριο συστατικό σήμανση ως προς την προέλευση. Το Συμβούλιο το απορρίπτει αυτό, δηλαδή δεν γίνονται τέτοια πράγματα για, συστατικά καθημερινά ή ε, εβδομαδιαία μπορεί να αλλάζει σε κατεργασμένα προϊόντα η προέλευση. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. Αλλά ποιο νόημα έχει για τον καταναλωτή αν μια επιχείρηση πουλάει ένα προϊόν κατεργασμένο και από το κύριο συστατικό να αναφέρει 20 πιθανές χώρες που αγοράζουν αυτό το βασικό συστατικό. Και αυτό γίνεται στην παγκόσμια αγορά, ξέρετε ότι είναι το εμπόριο παγκοσμιοποιημένο. Και τα κριτήρια για την αγορά είναι ε, η διαθεσιμότητα του συστατικού, η ποιότητα και η τιμή. Και βεβαίω μπορεί αυτό να διαφέρει από μέρα σε μέρα ή από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στη σήμανση και το επιχείρημα του Συμβουλίου Υπουργών. Για να φτάσουμε σε συμβιβασμό σε αυτό το σημείο όμως, νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες Κάπου αλλού που μπορούμε να βρούμε κάποια λύση είναι το θέμα της ετικέτας και του ευανάγνωστου. Δηλαδή, και εκεί συμφωνούμε, οι διαφορές μας είναι στο υποχρεωτικό ή όχι μέγεθος των χαρακτήρων, των γραμμάτων. 1,2 χιλιοστά το, το, το, το μικρό λέει το Συμβούλιο και είναι και μετακίνητο. Υπάρχουν προτάσεις κάποιων συναδέλφων να είναι ακόμα πιο μικροί οι χαρακτήρες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι επανάγνωστο και είμαι πρόθυμη να δεχτώ την πρόταση του Συμβουλίου 1,2 χιλιοστά. Αλλιώ, αν πάμε παρακάτω, είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Υπάρχει και πρόταση για 0,9 χιλιοστά, αλλά δεν ξέρω, όχι, είναι πολύ λίγο. Λοιπόν, Έχουμε και άλλες τροπολογίες που θέλουν ακριβώς το ίδιο, αλλά το λένε με διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετικά άρθρα. Και εκεί μπορούμε κάπως να ομαδοποιήσουμε και να συμφωνήσουμε. Παράδειγμα, η εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων έκανε τροπολογία η κυρία Τέισεν. Το είχα προτείνει και εγώ στην έκθεσή μου στη δεύτερη ανάγνωση. Ε, το προτείνουμε σε διαφορετικά άρθρα, αλλά εφόσον επιθυμούμε το ίδιο, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε που ταιριάζει καλύτερα σε ποιο άρθρο να μπει. Ένα τελευταίο πρόβλημα που θα ήθελα να σας αναφέρω και να το εξηγήσω, γιατί το θεωρώ πρόβλημα. Στην πρώτη ανάγνωση συμφωνήσαμε ε, ή ε, παραπέσεις απομιμήσεις τροφίμων να γράφονται. Το τυρί, ας πούμε, υπάρχει τυρί ε, από τυριού που είναι από, ζωικό, από φυτικό, λίπος. Αυτό είναι το γράφει, ότι δεν είναι τυρί, ότι είναι από τυριού. Το Συμβούλιο όμως τι λέει. Μα η απομίμηση καταρχήν δεν θα πρέπει να, δεν, να έχει το δικαίωμα να ονομάζεται τυρί να το λένε αλλιώ. Μόνο το σωστό τύρι λέγεται τύρι. Υπάρχουν κανόνε. Να γράψουμε, ξέρω εγώ, απομίμηση προϊόντο. Ε, λέει το Συμβούλιο Υπουργών ότι και αυτό είναι διφορούμενο. Το συζήτησαν ώρε ολόκληρε στην αντίστοιχη ομάδα εργασία και υπάρχει και κίνδυνο, το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα, να πει ένα κατασκευαστή στο τέλο ότι το δικό μου προϊόν δεν είναι απομίμηση, α, είναι καινοτόμο προϊόν. Είναι καινούριο, δεν απομιμείται ένα τυρί, είναι ένα άλλο προϊόν, καινοτόμο και νεωτερικό. Οπότε το Συμβούλιο Υπουργών τι προτείνει, όχι να μπει αυτή η λέξη απομίμηση στην πρόστια πλευρά. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξει και τις σκέψεις αυτές. Θα πρέπει να βρούμε κάποια κοινή λύση χωρίς να αναφέρουμε αυτή τη λέξη. Απομίμηση ή Πάντως και εκεί πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε. Προς το παρόν, σταματώ εδώ, εισαγωγικά ήθελα από αυτά. Θέλω να σας πω ότι για αύριο έχω συγκαλέσει τους σκιώδεις ηγητές συνεδρίαση για να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα και ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε βρει και αντίστοιχες διατυπώσεις για συμβαστικές τροπολογίες και να τις υποβάλω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις τώρα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τη συνάδελφο για την εξαιρετική της δουλειά. Η συζήτηση αυτή έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Όλοι νομίζω γνωρίζουν τι θα πει ο καθένας από εμά. Μου φαίνεται άσκοπο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση παρά τα αυτά γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, στη δεύτερη ανάγνωση αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να καλυφθούν οι ξεκάθαρες απαιτήσει του Κοινοβουλίου. Αυτές είναι σαφείς. Πολλά θέματα πρέπει να συζητηθούν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά. Πρώτον, τι θα πει ε, ε, το μπροστινό μέρος ε, θερμίδες, ε, λίπη, κορισμένα λίπη, σάχαρα, αλάτι, λέμε να είναι σε ένα σημείο, αλλά ποιο λένε ότι είναι αδύνατο να υπάρχουν, να υπά, ότι υπάρχει ε, να πούμε ότι υπάρχει μπροστινό μέρο της συσκευασία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ανοησία. Υπάρχει σαφή ε, ε, μπροστινή πλευρά. Υπάρχουν θρεπτικέ ουσίε στα τρόφιμα και όταν είναι σαφώς αναγεγραμμένα στο μπροστινό μέρο της συσκευασία δεν χρειάζεται ε, να κουραστεί πολύ ο καταναλωτής για να ενημερωθεί για αυτά που θέλει. Πρέπει να είναι σαφές και στο μπροστινό μέρος. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα παθήσεις όπως η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος και ο διαβήτης, πρέπει οι καταναλωτές να μπορούν να γνωρίζουν ότι υπάρχει η υπάρχουν οι απαραίτητε πληροφορίε για να κάνουν υγιεί επιλογέ αν το επιθυμούν. Ο καταναλωτή θέλει αυτέ τι πληροφορίε, Το κοινοβούλιο τη ζητά και επ' αυτού δεν είμαι διατεθειμένη να συμβιβαστώ. Τώρα, όσον αφορά την χώρα προέλευση, το κοινοβούλιο ήταν απόλυτα σαφέ ότι θέλουν να είναι υποχρεωτική αυτή η προέλευση, κυρίω για το κρέα. Η θέση του Συμβουλίου είναι ότι υπάρχει επισήμανση στα προϊόντα κρέατος θα δουν το θέμα της προέλευσης για τα ε, γαλακτοκομικά και άλλα σε πέντε χρόνια. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η υποχρέωση για το κρέας, αλλά πρέπει άμεσα να ε, συμπεριληφθεί και το κρέας σε ε, επεξεργασμένα προϊόντα. Δεν νομίζω ότι πρέπει γι' αυτό να περιμένουν πέντε χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένουν καταναλωτές ότι ένα προϊόν είναι ας πούμε ένα σάντουιτς με κοτόπουλο να είναι αγγλικό ενώ το ε, κρέας έρχεται από την Ταϊλάνδη. Ε, μπορούν να πούν ασαφής προέλευση ή απροσδιόριστη. Αλλά οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν από πού προέρχονται τα τρόφιμά τους και έχουν και το δικαίωμα να το γνωρίζουν. Αυτό νομίζω είναι σοβαρό ζήτημα. Τέλος, θέλω να επικεντρωθούμε σε, αυτό, σε αυτά τα Λύπη τρανς που συνδέονται με Αλσχάιμερ, με καρδιοπάθειες, με ε, περιορισμένη γονιμότητα και εδώ το Συμβούλιο μιλάει για εθελοντική επισήμανση. Δεν το ξέρω. Αν υπάρχει εθελοντική επισήμανση για ε, αυτά τα λιπαρά, τα τρανς, αν πάρει κάποιος δύο προϊόντα που, περιέχουν και τα δύο, το ένα λέει ότι έχει και το άλλο δεν έχει, αυτός ο καταναλωτής θα θεωρήσει ότι αυτό που δεν αναφέρει θα ε, είναι το υγιέστερο. Είναι πάρα πολύ παραπλανητική αυτή η επιλογή και δεν νομίζω ότι πρέπει να την επιτρέψουμε. Θα ήθελα ε, να ε, να απαγορευτούν αυτά. Ας το συζητήσουμε. Η Δανία το επέβαλε. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν είμαι υπέρ καθόλου της εθελοντικής επισήμανσης για τα λιπαρά τρανς. Αυτό είναι εξαιρετικά παραπλανητικό. Αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι νομοθεσία για ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Πρέπει στο επίκεντρο να βρίσκεται αυτό που επιθυμούν και αυτό που χρειάζονται οι καταναλωτές, σαφώς. Και πρέπει να σκεφτούμε τα τεράστια ωφέλη για τη δημόσια υγεία που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη νομοθεσία. Η επισήμανση πρέπει να είναι εύληπτη, πρέπει να είναι έντιμη, να μην είναι παραπλανητική και να υπάρχει για να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές που θέλουν. Άρα υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα τα οποία δεν θα πρέπει καν να τα συζητάμε ε, ε, με, ε, με σκοπό τη συμβιβαστική λύση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που με ανησυχούν εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν, δεν είναι στην αίθουσα εμφανιστούν, θα του δώσουμε το λόγο. Θα περάσουμε λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι γενικά ε, για τις τροπολογίες. Παραμένει υπερβολικός ο αριθμός τους. 402 τροπολογίες για δεύτερη ανάγνωση ε, σε επιτροπή είναι πάρα πολλές. Δεν είμαι καθόλου βέβαιη αν θα καταφέρουμε να βρούμε λογικές συμβιβαστικές προτάσεις, θα δείξει. Ε, είπε η κυρία Βίλμον πάρα πολύ λογικά πράγματα. Εγώ να μιλήσω μόνο για τις δικές μου τροπολογίες. Η χώρα προέλευσης πρώτα. Κάναμε τις τροπολογίες αυτές και σε πρώτη ανάγνωση, τις εγκρίναμε και τώρα έχουν κατατεθεί πάρα πολλές διαφορετικές για αυτό το θέμα. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η ενημέρωση, η πληροφορία για το πόθεν έρχεται ένα προϊόν ή το βασικό του συστήμα. Θέλουν και προδείξουν. Δεν ξέρω. τα Πάρα πολλά την καθημερινή ανθρώπους να μου λένε ότι αυτό θέλουν από εμά Έχουν αλλάξει οι καιροί, έχουν εξελιχθεί. Και πρέπει να υποχρεωτικά να ομολογήσω κι εγώ ότι και η συγκήτρια... Τι έγινε, υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία στα αγγλικά. Υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία. Είπε ε, ότι υπάρχει πρόβλημα στη συζήτηση στο Συμβούλιο. Κοιτάξτε, εμένα δεν με εντυπωσιάζουν αυτά. Θα πάμε στη συνδιαλλαγή. Γιατί νομίζω ότι θα πάμε στη συνδιαλλαγή, γιατί σε δεύτερη ανάγνωση δεν πιστεύω να έχουμε συμφωνία. Ε, αν δούμε πώ έχουν οι τροπολογίε και η προθυμία ε, γενικότερα. Αν μπούμε στη θέση των παραγωγών, που είναι και αυτή σημαντική. Ε, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε, είναι εφικτό αυτό και για τους παραγωγούς. Ε, τότε θα βρούμε μια ε, λύση συμβιβαστική. Τα μεμονωμένα προϊόντα θα πρέπει να γράφουν τι είναι. Ε, ε, όχι μόνο το κρέας βεβαίως, όλα τα ζωικά προϊόντα, γαλακτοκομικά και τέτοια που είναι ένα προϊόν, ένα συστατικό και για τα άλλα προϊόντα που έχουν ένα βασικό συστατικό νομίζω ότι μπορούν να επισημένονται και μιλώ για υποχρεωτική σήμαση, εδώ, προσέξτε, όπως έλεγε ο συμβιβασμό μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείε που έχουν συμβάσεις με 20 τουλάχιστον χώρες ή παραπάνω. Ναι, το ξέρω ότι υπάρχουν. Παράδειγμα, από τη Γερμανία. Ξέρω ότι υπάρχουν κατασκευαστές που βγάζουν ένα γλύκισμα, α πούμε, και χρειάζονται αμύγδαλα. Ναι, το πιστεύω ότι εισάγουν από διαφορετικές χώρες, αλλά όχι και 20. Μπορεί να είναι 4 ή 5 οι προμηθεύτριε χώρες αμυγδάλα. Και ε, όπως και για τα ψάρια, α πούμε, μάλλον και για τις νοπές συσκευασίε. αυτό λύνεται. Ε, θέλω να καταλάβει ο, κλάδος ότι τον καταναλωτή ε, τον ενδιαφέρει και θέλει να κάνει μια προσπάθεια. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή την προσπάθεια από την πλευρά της βιομηχανίας και με ενοχλεί αυτό. Το ίδιο ισχύει και για ε, τις θερμίδες ε, και για τις μερίδες. Ανέκαθεν πίστευα ότι Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και πάρα πολύ πρόθυμοι να λέμε ε, στους κατασκευαστές ποια είναι η μερίδα. Μα κοιτάξτε, συνήθως είναι ένα κουτάλι, μια φέτα, ένα φλιτζάνι, ξέρω εγώ, αυτό περιμένω να γράφει. Και αυτό θέλουν οι καταναλωτές, θέλουν να ξέρουν ποια είναι η μερίδα. Όχι να κάθονται, να κάνουν μέθοδο των τριών, να ε, βρίσκουν, ξέρω εγώ, να ζυγίσουν το μουσλι, να δούνε πόσα γραμμάρια είναι και πόσε θερμίδε θα φάνε ή να βγάλουν κουταλιέ, ξέρω εγώ. Δεν τα θέλουν αυτά οι καταναλωτέ, θέλουν ξεκάθαρα, σταρά τα λόγια και μπορεί να το κάνει αυτό η βιομηχανία. Δεν είμαι καθόλου πρόθυμη για συμβιβασμό εκεί για το μέγεθο τη Μερίδα. Και ούτε εθελοντικά σε καμία περίπτωση υποχρεωτικά να γράφουν ποια είναι η θερμίδα, πώ την επιλέγουν και πόσο. Αυτά. Και τέλος, για ένα θέμα που συζητήσαμε στην αρχή και είναι δική μου η τροπολογία, 392 με του κυρίου Κράμε, αυτό που είπαμε στην αρχή και το είπε και η κυρία Μακάβαν, ότι έρχονται εδώ πέρα τα λόμπι και μας βάζουν έγγραφα στο γραφείο γιατί πιστεύουν ότι δεν διαβάζουμε τα mail μας. Το είπα και προηγουμένως όταν ήμασταν λιγότερο εδώ ότι δεν εξυπηρετεί αυτό και θα φροντίσω στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου που έχουμε ε, νέα ομάδα για τη διαφάνεια να τους δυσκολέψω την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι υπηρεσία αυτό, δεν είναι καλή ιδέα και εκείνοι από τους πελάτες τους και μεμονωμένους παρασκευαστές θα το ε, μετανιώσουν και ελπίζω να ε, σας τιμωρήσουν γι' αυτό. Επίσης μιλήσαμε και για χρωστικές ουσίες. Η κυρία Ζόμερ είχε κάνει μια αρχική τροπολογία για ε, χρωστικές ουσίες στο τρόφιμα και αυτή η τροπολογία προβλέπει στο παράρτημα ε, που αναγράφονται αυτά ε, τα τρόφιμα και συγκεκριμένα στο παράρτημα 7β και ο ρυθμός 15α νέο να προβλέπει βέβαια ότι όταν είναι, φρούτα, λαχανικά, φυτά κτλ. Είναι, μπορεί να είναι χρωστικές ουσίες μετά από ειδική επεξεργασία, κατεργασία και να γράφει ότι είναι τρόφιμα αυτές οι χρωστικές. Και κανέναν δεν θα εκπλήξει ότι ας πούμε ένα παντζάρι, ένα σπανάκι, ένα καρότο που έχει χρώμα είναι άλλο πράγμα ως χρωστική ουσία και άλλο είναι χημική ουσία που του βάζεις για να χρωματίσει το τρόφιμα. Και για ποιο λόγο τώρα θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη χάρη σε κάποιο κλάδο ο οποίος παράγει χημικά ε, προϊόντα, ουσίες για να χρωματίζονται ε, τρόφιμα και να τιμωρήσουμε εκείνον που χρησιμοποιεί μόνο φυτικές ε, ουσίες για χρωματισμό των τροφίμων. Γι' αυτό έκανα αυτή την τροπολογία για να επανέλθει η κατάσταση της πρώτης ανάγνωσης, η κυρία Σόμερ δεν επανέλαβε την τροπολογία της. Ελπίζω να την υποστηρίξει και σε δεύτερη ανάγνωση. Από κοινού την υποβάλαμε, γιατί είμαι πεπισμένη ότι είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Γιατί αυτό είναι τρόφιμα που βάφουν άλλα τρόφιμα και θα πρέπει να το πούμε. Δεν είναι χρωστικές ουσίες, συμβατικές, χημικές, ε, κατασκευασμένες. Γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αυτό έκανα κι εγώ. Αυτές τις τροπολογίες περιορίστηκα, ξέρω ότι υπάρχουν άλλοι και άλλες τροπολογίες. Για μένα αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι και σημεία κλειδιά για οποιαδήποτε προσπάθεια συμβιβασμού. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω για τρία ζητήματα, στα γρήγορα. Πρώτον, για το ευανάγνωστο όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος των, της ετικέτας. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε ότι μας κατέβει στους ε, επιχειρηματίες. Το έχουμε συζητήσει και πήραμε υπεύθυνη απόφαση ε, επιβάζοντας, ε, καταργώντας το, με ελάχιστο μέγεθος. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν το επιθύμησε. Γι' αυτό με τον συνάδελφο ε, υποβάλαμε τροπολογίες να περιοριστεί ε, το μέγεθος αυτό στο ένα χιλιοστό για να μην ε, τιμωρούνται αυτοί που έχουν τις μικρότερες συσκευασίες. Είναι επικίνδυνο για συγκεκριμένα πρόγραμματα, ελάχιστα μεγέθη όσον αφορά τις ρεπτικές ουσίες γιατί έτσι κι αλλιώς ε, υπάρχει ιδιαίτερη νομοθεσία για αυτά τα ε, προϊόντα και αυτό είπα στην ε, τροπολογία 171. Πρέπει το να αυξηθεί ο όγκος ή το μέγεθος για να υπάρχουν οι πληροφορίες, κινδυνεύουμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο θα παραμείνει, δεν θα καταναλωθεί και θα ε, διατηρείται σε ακατάλληλες ε, συνθήκες ή σε υπερβολικά μεγάλη διάρκεια και αυτό για κάποιους πληθυσμούς, ευαίσθητες ομάδες μπορεί να είναι επικίνδυνο. Τώρα όσον αφορά την προέλευση, πολύ λεπτό το ζήτημα, γιατί ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πολίτες μας που θέλουν να γνωρίζουν την προέλευση κάποιων προϊόντων. Γι' αυτό έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες που αναφέρουν υποχρεωτικά την προέθελευση των συστατικών που μπαίνουν σε ένα προϊόν όταν μιλάμε για ποσότητες που πλησιάζουν το 50%. Είναι νομίζω σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές για την προέλευση των βασικών συστατικών των τροφίμων τα συστατικά αυτά ε, έχουν συσχετιστεί από τον καταναλωτή με το τρόφιμο και θα είναι αυτά που φτάνουν περίπου το 50%. Όταν είναι βεβαίως η προέλευση διαφορετική από αυτή που ε, αναφέρεται για το τρόφιμο. Είναι σημαντικό αυτό γιατί θεωρώ ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την προέλευση των σημαντικών συστατικών των τροφίμων. Τώρα, όσον αφορά το αλάτι. Με τις συναδέλφους μου στο, στην τροπολογία, βάλαμε το 232, την τροπολογία 232 είναι σημαντικό ε, έχει και άλλες τροπολογίες. Το αλάτι αυτό, ε, το νάτριο αυτό, με συγχωρείτε, υπάρχει ε, φυσικά σε τρόφιμα που δεν έχουν αλάτι, όπως το γιαούρτι και το γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να γνωρίζει την πραγματική περιεκτικότητα του νατρίου στο, ε, στα τρόφιμα και πρέπει λοιπόν ο παραγωγός να διευκρινίσει και να συμπληρώσει τις υποχρεωτικές πληροφορίες που αφορούν το αλάτι. Αυτά ήταν τα σημεία στα οποία ήθελα συγκεκριμένα να παρέμβω. Ευχαριστώ κυρία Κράμαρ. Ευχαριστώ και εγώ σύντομος θα είμαι. Αρχίζω από την προέλευση και τη σήμανση αυτή και θα ήθελα να μπω ε, σε αυτό που είπε η κυρία Ροτ Την τιμά αυτό να ενημερώνονται όσο γίνεται περισσότερο ε, για την προέλευση του προϊόντος οι καταναλωτές, προϊόν που αγοράζουν και στη συνέχεια θα φάνε. Αλλά πιστεύω ότι το Συμβούλιο έχει επιλέξει τη σωστή προσέγγιση που λέει χωρίς αντίκτυπο, χωρίς μελέτη αντικτύπου, χωρίς μελέτη επιπτώσεων δεν είναι τόσο εύκολο. Και η κυρία Ροτμπέρεντ είπε ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στους καταναλωτές. Ε, είναι πολύ γρήγορο το πούμε. Κοιτάξτε, το κέτσαπ, ντομάτας ή το γιαούρτι το θέμα δεν είναι ότι έρχονται από 20 διαφορετικέ χώρε οι ντομάτε ή το γάλα, αλλά θέλουμε να βρούμε συμβιβασμό. Θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε μέχρι πού θα υποχρεώνουμε ε, την αναγραφή της προέλευση. Γιατί και εγώ είμαι επιχειρηματίας και μπορεί να σας πει ένας επιχειρηματίας ότι είναι και θέμα κόστος από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει την ετικέτα για την επόμενη παρτίδα ε, του κέτσαπ που θα ε, παράγει. Ε, και υπάρχουν πολλά προϊόντα, σας έδωσα δύο παραδείγματα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πόσο χρήσιμη στο κάτω-κάτω είναι η τελική ενημέρωση του καταναλωτή. Να μην καούν λοιπόν τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Για τα κατεργασμένα προϊόντα ή μεταποιημένα που πάνω από 50% ε, έχουν ένα συστατικό, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει μελέτη αντικτύπου ή να πούμε με την επιφύλαξη ότι θα γίνει τέτοια μελέτη. Και κόστος ωφέλους. Και βεβαίως υπάρχουν προϊόντα όπου ενδιαφέρονται και οι ίδιοι οι, ε, παρασκευαστές να το κάνουν ας πούμε γιατί είναι ένα ε, προϊόν τοπικό και χαρακτηριστικό ας πούμε ε, τα, το τουρσί, τα αγκουράκια Σπρέβαλτ στη Γερμανία ε, είναι ένα προϊόν με σήμα κατατεθένες που το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Τώρα, έχουμε μια πολύ ακαδημαϊκή συζήτηση για το πού θα πρέπει να μπαίνουν αυτές οι ενδείξεις. Έχει νόημα αυτό που λέει το Συμβούλιο. Έχει σημασία η σκοπιά. Από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς και να φαίνεται και όχι να γράφει ο νόμος που ακριβώς πρέπει να αναγράφεται αυτό πάνω στη συσκευασία. Είναι εύκολο να πάρεις από το ράφι, εν περιπτώσει, στο χέρι σου το προϊόν, να το γυρίσεις από την πίσω μεριά και να το διαβάσεις. Είναι ανάγκη να είναι μπροστά και είναι και πολύ ιδεολογική ε, η συζήτηση αν θα πρέπει όλα οπωσδήποτε να αναγράφονται στην πρόσθεια πλευρά. Να είναι εμφανές, ανάγνωστο το μήνυμα στην ετικέτα και θα το βρει ο καταναλωτής. Στο μεταξύ τρία χρόνια το συζητάμε αυτό το θέμα. Ε, ως κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να σκεφτούμε και την ενιαία αγορά. Είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτή της, ε, της πρότασης και στην πρώτη ανάγνωση το είχαμε πει, ότι οι ε, εθνικές ρυθμίσεις έκτακτες πρέπει να είναι προσθήκη στα όσα λέμε τώρα εδώ. Ε, αλλά να γίνει όσο γίνεται περιορισμένες, γιατί πρόκειται για εσωτερική αγορά, για μια ελάχιστη εναρμόνιση. Τώρα αν έρχονται τα κράτη-μέλη ε, να κάνουν δικές τους ρυθμίσεις πέρα από τα όσα εμείς εδώ αποφασίζουμε, χάνουμε το σκοπό μας και ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν τους εκπροσωπούν λόμπι και είναι πολλές στην παραγωγή τροφίμων δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Πέρα από τον κανονισμό μας δηλαδή αν βάλουν οι χώρες επιπλέον νομοθεσία. Και για αυτές τις ε, φυτικές βαφές ας πούμε χρωστικές ουσίες ε, τα είπε η κυρία Ροτμπέρντ με καλούν και εμένα διάφοροι και με ρωτάνε σύνδεσμοι και ενώσει παραγωγών πώ θα εκπροσωπούνται καλύτερα στο κοινοβούλιο, να σα πω πώ δεν πρέπει να γίνεται έτσι όπω μα βάζει τα έγγραφα σήμερα στα έδρανα. Αυτό αποκλείεται. Και ε, ε, αμέσω πριν την ψηφοφορία που έτσι κι αλλιώ δεν γίνεται και έχουμε και 400 τροπολογίε να παίρνουμε χαρτιά πάνω στα έδρανα στην Επιτροπή. Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό παράδειγμα ακριβώς για το τι δεν πρέπει να κάνουν οι εταιρείε. Αφήστε δε που οι ισχυρισμοί επίση είναι ψευδοί και λαθασμένοι και εγώ τις αμφισβητώ. Τι λέει εδώ ότι στο μέλλον θα μπορούν να χρησιμοποιούν ό,τι θέλουν οι κατασκευαστές ε, χρωστικών από οποιαδήποτε φυτά. Αυτά είναι θράσος, είναι πραγματικά σκέτη ανέδεια που γράφουν. Εδώ μιλάμε για ισχυρισμούς, όχι για ε, την νομοθεσία για τα πρόσθετα. Άλλο πράγμα συζητάμε, όχι, ε, τι θα γράφει ετικέτα. Είναι ε, θράσος είναι ε, ανέδεια ε, στο τετράγωνο και έχω πολλά να πω, αλλά αν θέλετε εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο, αυτό είναι ο χείριστος τρόπος για να γίνει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έμπνερ. όχι, συγγνώμη. Η κυρία Χιούμπνερ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι η ενημέρωση θα πρέπει να εξυπηρετεί τον Ευρωπαίο πολίτη και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται μας κατευθύνουν μόνο ε, τα λόμπι. Όσον αφορά τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για πολλές ε, πληροφορίες που προτάσουν και τα λόμπι. Τώρα, εγώ συμβουλεύτηκα το αρμόδιο Ινστιτούτο της χώρας μου και με βάση τα όσα κατάλαβα έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε καταρχήν την ακαδημαϊκή έρευνα. Για τις τροπολογίες με τη χώρα προέλευσης δεν συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους εδώ και δεν συμφωνώ με την ιδέα ότι ορισμένες πληροφορίες είναι δύσκολο να κατανοηθούν, ιδιαίτερα για τα κύρια συστατικά που πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς αν ε, το συστατικά προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, αν το κρέας είναι από τη Λατινική Αμερική και ε, δεν μας βοηθά το να μην έχουμε πληροφορίες ε, ας πούμε για το αν ένα προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Πρόσφατα αγόρασα σκόρδο και προερχόταν από την Ισπανία. Μα φτιάχνουν δύο είδη. Μάλλον πουλούσαν δύο είδη σκόρδου. Το ένα ήταν από την Ισπανία, το άλλο ήταν από την Κίνα. Πολύ σημαντικό να έχουμε τις πληροφορίες στην μπροστινή πλευρά της συσκευασία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την προέλευση, εντάξει. Αλλά αν κανείς δεν μπορεί να διαβάσει τα γράμματα γιατί είναι τόσο μικρά ή γιατί το πίσω μέρος είναι χρωμα... μάλλον το... η βάση είναι σε τέτοιο χρώμα που να μην μπορείς να τα διαβάσεις δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Δεν πρόκειται κανείς να πάει στο σούπερ μάρκετ με μεγεθυντικό φακό για να διαβάσει πληροφορίες Αν δεν είναι βανάγνωστο, δεν είναι βανάγνωστο. Και δεν αφορά μόνο το μέγεθος μέγεθο τη γραμματοσυρά, αλλά και το φόντο, το χρώμα του φόντου. Και εδώ υπάρχουν ε, δυνατότητες όσον αφορά την ενεργειακή αξία του προϊόντος. Αν πρόκειται για προσκευασμένο προϊόν, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί που εγώ, από εκεί που προέρχομαι, πολύ λίγοι κουβαλάνε μαζί τους υπολογιστή για ε, κομπιουτεράκι για να υπολογίζουν ε, <laughs> την... Ε, τις θερμίδες. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να τρώνε χαμηλά λιπαρά γιατί έχουν προβλήματα υγείας. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν αν αναγράφεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο να βοηθήσουμε τους διαβητικούς ή τους ανθρώπους που υποφέρουν από αλλεργίες. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Να ξέρουμε επίσης ποια είναι η μερίδα Και αν στην προστινή πλευρά λέει ότι 100 γραμμάρια ε, ε, σημαίνει τόσες θερμίδες, ενώ από την πίσω πλευρά λέει ότι το πακέτο περιέχει 125 γραμμάρια, κανείς δεν θα κοιτάξει την πίσω πλευρά και να υπολογίσει ακριβώς πόσες θερμίδες έχει αυτό το προϊόν. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτές οι πληροφορίες είναι λίγο παραπλανητικές και θα πρέπει να βρούμε μια πιο πρακτική προσέγγιση. Θα πρέπει να μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει και ακόμα και αυτοί που έχουν πραγματικά χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες. Ο κύριος Κυλακάκης. τα ακούγε μόνος του. Uh, λοιπόν, δύο θέματα θέλω να θίξω. Η χώρα προέλευσης. Αυτή ενδιαφέρει τους καταναλωτές μαθαίνουν πολλά πράγματα για το προϊόν με πολύ απλό τρόπο που δεν μπορούν να μάθουν με κανέναν άλλο τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά έχουμε ένα ε, πάθος, ένα φοβερό ενδιαφέρον για τη χώρα προέλευσης και πρέπει το σεβασμό, να σεβαστούμε αυτή τη στάση των καταναλωτών και ψηφοφόρων. Συμφωνώ ότι χρειάζεται μελέτη επιπτώσεων, όμως εγώ θα έλεγα ότι προηγούνται οι καταναλωτές από τους παραγωγούς στην προκειμένη περίπτωση, από τους κατασκευαστές. Τελικά, εμείς παράγουμε, η παραγωγή γίνεται υπέρ των καταναλωτών. Δεύτερον, μια τροπολογία που είχε ψηφιστεί ως αιτιολογική σκέψη στην πρώτη ανάγνωση για τα, τους κινηματογράφους multiplex που προσφέρουν κάποιο είδους διατροφικές πληροφορίες στα επιτόπου συσκευασμένα τρόφιμα που παράγουν. Μιλάμε για μη σκόπιμα γεύματα με ελάχιστη και αρνητική θρεπτική αξία της τάξεως των 500 έως 1000 θερμίδων και εκατομμύρια θα έλεγα νέοι τα αγοράζουν αναψυκτικά, οι popcorn που δεν έχουν την παραμικρή διατροφική πληροφορία. Είναι ένα γεύμα που δεν σκόπευαν να το πάρουν και δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι ακριβώς κάνουν. Δεν υπάρχει παραμικρή πληροφορία. Σε ένα, μια περίοδο που υπάρχει επιδημία παχυσαρκίας ε, των εφήβων στην Ευρώπη, και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Θεωρώ ότι η τροπολογία αυτή είναι σημαντική, η οποία θα αλλάξει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ελπίζω ότι θα ξεπεράσουμε... Δεν είναι σκοτεινά στο κινηματογράφο. Όχι. Αυτοί που πηγαίνουν σε αυτούς τους κινηματογράφους ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ φωτεινά στο χώρο που παίρνεις το που αγοράζεις αυτό που θα φας. Στα σκοτεινά το τρως, αλλά εκεί που τα αγοράζεις έχει φως. Συζητάμε για καθαρές θερμίδες, γεμάτες ακόρεστα λίπη και ζάχαρη. Ποπκόρν, αναψυκτικά δεν προσφέρουν τίποτα άλλο παρά ζάχαρα, ε, άμυλο και, και κορεσμένα λίπη. Τίποτα άλλο. Και τα παίρνουν νέα παιδιά δεκάδες εκατομμύρια νέα παιδιά που δεν έχουν κανέναν τρόπο να μάθουν τι ακριβώς τρώνε. Και βεβαίως οι γονείς τους δεν είναι εκεί. Πολλοί από αυτούς είναι έφηβοι, πολλοί είναι νέοι οικοσάριδες που αυτοί είναι εξάλλου αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν σε τέτοιου είδους κινηματογράφους, τα multiplex. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεραστούν οι τυπικές δυσκολίες και να υπερψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ κύριο Ρώση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν Διαπιστώνουμε πως η συγχύτρια σε ορισμένα πράγματα έχει ανταποκριθεί σε κάποια από αυτά που εγώ είχα προτείνει. Όμως υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία που είναι αντίθετα, όπως ας πούμε η υπόδειξη για το ενεργειακό περιεχόμενο σε ανά 100 γραμμάρια. Αυτό πολύ συχνά γιατί ως, στο, στο λάδι ας πούμε ή σε προϊόντα πολύ Ε, με πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες όπως στο λάδι ας πούμε η περίφημη αυτή δόση ε, είναι ένα κουτάλι της σούπας 100 ε, γραμμάρια λάδι είναι 900 θερμίδες εναντί των 80 ή 90 που βάζει κανείς στο φαγητό του να συνεχίζουμε να επιμένουμε λοιπόν για τα 100 γραμμάρια σημαίνει ότι τελικά δεν βοηθάμε τον καταναλωτή. Τουλάχιστον όταν θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτή την ένδειξη που είναι κατά τη γνώμη μου περιττή και πλονασματική, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να βάζουμε τα 100 γραμμάρια ή δόση ή μερίδα και τις, ή και τις δύο ενδείξεις, γιατί πραγματικά διαφορετικά η κατάσταση είναι γελία. Τώρα, όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων και των συστατικών, οπωσδήποτε θα πρέπει να μπαίνουν. Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε για το συμφέρον ε, των καταναλωτών και ότι είναι ντροπή ε, τα όσα ζητάνε τα λόμπι, μα οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν τι τρώνε. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην λέμε από πού έρχεται το προϊόν και τα συστατικά του. Φοβόμαστε να μιλήσουμε για λανθασμένα συμφέροντα για ορισμένε εταιρείε. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να λέμε από πού προέρχονται τα αισθητικά. Τι φοβάστε, τι φοβάστε. Θα πρέπει να λέτε από πού προέρχεται το κάθε προϊόν. Άμα θέλουμε να, μιλάμε ότι είμαστε, να λέμε ότι είμαστε υπέρ του καταναλωτή, θα πρέπει να λέμε από πού προέρχονται τα συστατικά. Τώρα, για το φανάρι. Ε, εγώ είμαι ικανοποιημένο για τι τροπολογίε Τη 40 στην, στο άρθρο 9 και την 77 στο άρθρο 34, γιατί αφαιρούμε μια σχέδια διαπαντό τη δυνατότητα να ανατρέχει κανεί σε υποδείξει που είναι περιττέ. Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο επικίνδυνη μια διαιτητική ζάχαρη σε σχέση με ένα προϊόν όπω το σαλάμι ή το τυρί, γιατί έχουν, που έχουν όντω υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Δηλαδή το να βλέπεις ένα τυρί με ένα κόκκινο φανάρι, σπρώχνει τον καταναλωτή να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο προϊόν και όχι το τυρί. Το άλλο προϊόν όμω μπορεί να τον βλάψει περισσότερο. Εντάξει, δεν τρώει κανεί ένα κιλό τυρί γιατί θα του πονέσει κοιλιά. Άμα όμω ε, φάει κανεί ένα κιλό μαϊδανό πάλι θα του πονέσει η κοιλιά του. Ή αν φάει ένα κιλό φύλλα δάφνη, τα ίδια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε ένα κιλό μαϊντανός έχει πολύ λιγότερες θερμίδες από ένα κιλό τυρί. Παρ' όλα αυτά προκαλεί πονόκυλο. Τα βασικά προϊόντα θα πρέπει λοιπόν να πολλούνται με διάφορες γλώσσες της ένδειξης, δηλαδή να είναι μεταφρασμένα. Πολλά πολλούνται στα αεροδρόμια. Πολλά προϊόντα πολλούνται σε δομή. Γιατί λοιπόν αυτό που κατασκευάζει το προϊόν δεν μπορεί να τα γράφει σε διάφορε γλώσσε. Και μάλιστα να απαγορεύουμε και τη χρήση των πολλών γλωσσών. Εγώ θα ήθελα να μπορώ να καταλάβω και τα αγγλικά, ναι, εντάξει, υποχρέωση για τα αγγλικά. Αλλά γιατί ο παραγωγός να μην μπορεί να τα γράφει και στα Ιταλικά ή στα Γαλλικά, άμα ο παραγωγός είναι Ιταλός ή Γάλλος, ή στα Γερμανικά, άμα είναι Γερμανός. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διάταξη. 32 β νέο. Τροπολογία 32 β νέα. Και εδώ κάτι πολύ παράξενο. Παρεμβαίνουμε απαγορεύοντας τη δημοσίευση μείωσης της ζάχαρης και των λιπαρών. Ακόμα και αν δεν μειώνονται ταυτόχρονα οι θερμίδες. Και εδώ ρωτώ τους πράσινους να που συνήθως τα ξέρουν αυτά. Αν εγώ όμως μπορώ να υποκαταστήσω τη ζάχαρη και τα λιπαρά, και ίσως προσθέτοντας ε, ίνες, που οι ίνες έχουν πολλές ε, θερμίδες, αλλά που είναι θερμίδες που τις ε, απορροφά άμεσα το σώμα μας. Άρα δεν προκαλούν καμία ζημιά, αντιθέτως κάνουν καλό. Αν μπορώ λοιπόν να αφαιρέσω τα λιπαρά και τις ζάχαρες, για τα ζάχαρα, γιατί δεν μπορώ να το πω, αφού οι ίνες κάνουν καλό και εγώ καταφέρνω να αντικαταστήσω τα ζάχαρα και τα λιπαρά προσθέτοντας ένα ποσοστό ινών. Οι θερμίδες είναι οι ίδιες, αλλά δεν μπορώ να το αναφέρω. Και αυτό είναι μυστήριο. Α, τώρα, αν, αναγνωσιμότητα, ανάγνωστος χαρακτήρας δηλαδή των γραμμάτων πάνω στις συσκευασίες. Τώρα, α, οποιοδήποτε πράγμα αλλάξει και πρέπει να τροποποιηθεί, θα πρέπει να επανέλθουμε και να ψηφίζουμε το κείμενο αυτό στην Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, αλλά αυτό είναι παράλογο. Καλύτερα είναι να τα αναθέσουμε αυτά στην Κομισιόν, όπου υπάρχουν τεχνικοί που μπορούν να αξιολογήσουν ποια είναι τα πιο κατάλληλα μέτρα και που διαπιστώνουν ότι αν ε, είναι λάθος επανέλθουν εκεί και θα διορθωθούν. Όχι να έρχονται ξανά όλα στο Κοινοβούλιο. 66 σελίδα 38, τροπολογία 68. Σελίδα 38. Και εδώ, η Ενδείξεις οι θερμιδικές συνδέονται με την ημερήσια ανάγκη σε θερμίδες μιας μέση γυναίκα, μέσης ηλικία. Όλοι ξέρουν ότι οι θερμίδες είναι διαφορετικές για γυναίκες και άντρες. Ε, περίπου 500 θερμίδες διαφορά. Μια ενήλικη γυναίκα μέσης ηλικία, ε, αν, αν ο άντρας καταναλώσει αυτά στις θερμίδες θα πεθάνει της πείνας και άσε που έχουν για διαφορετικά χαρακτηριστικά άντρες, γυναίκε, παιδιά, γέροι κτλ. Α βγάλουμε έναν μέσο όρο. Ένα μέσο όρο για τη γυναίκα, ένα μέσο όρο για τον άντρα. Τα βάζουμε στη μέση, τα διαιρούμε δια δύο. Άρα δηλαδή 2.000 και 2.500 θερμίδε μα κάνει 2.050. Ε, δεν μπορεί να λέμε για όλου το ίδιο. Δίνουμε μία προσέγγιση. Διαφορετικά είναι γελίο αυτό που κάνουμε και είναι παραπλανητικό για το υπόλοιπο ίμιση του κόσμου, αν πάρουμε ως βάση μόνο τη γυναίκα. Κάτι ακόμα τώρα που δεν έχει επιληθεί. Πρέπει η συγκήτρια να μου εξηγήσει όταν έχουμε μία σούπα μινεστρών κατεψυγμένη ή ένα μίξ ε, ψαριών με 10-12 διαφορετικά ψάρια και 14 διαφορετικά λαχανικά κατεψυγμένα, πώς είναι δυνατόν να υποδειχθεί η ημερομηνία κατάψυξης, γιατί το κάθε κομμάτι σε αυτό το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει καταψυχθεί σε διαφορετική στιγμή. Ο κάθε ψαράς ε, τα καταψύχει με το που φτάνουν στην γη ή ακόμα και μέσα στο σκάφος του. Μετά τα βάζει σε μεγάλα κοντέινερ, τα ανακατεύουν με 10 διαφορετικά είδη ψαριών και σε ένα άλλο κοντέινερ 10 διαφορετικά είδη λαχανικών. Ε, πώς θα γράψουμε και τι ημερομηνία θα γράψουμε. Τι θα δει δηλαδή 18 διαφορετικές ημερομηνίες κατάψυξης ενώ θεωρητικά η και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος θα είναι 18 διαφορετικές ε, ημερομηνίε. Δηλαδή, άλλη ημερομηνία λήξης για το μαϊντανό, άλλη για το καρότο, άλλο για, το πατά, για την πατάτα. Και ε, καλύτερα να βάζουμε και ένα βιβλίο λοιπόν ε, δίπλα στο, προϊόντο, στο προϊόν να λέει ας πούμε ότι τα φασόλια λήγουν σε 6 μήνες, τα καρότα σε 3. Τώρα, στη σελίδα 17 έχουμε και εδώ τονίσει ένα πρόβλημα, γιατί άλλο είναι η ημερομηνία όπου έχει συσκευαστεί το σαλάμι, το κόβουν σε φέτες και το δίνει στον πελάτη φρέσκο ας πούμε, στην πρώτη περίπτωση ότι δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί ο κανόνας της ετικετοθεσίας γιατί το κόβω και το δίνω στον πελάτη κατευθείαν. Ενώ όταν το κόβω, το συσκευάζω αριστογός και το βάζω στο ράφι είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Επίσης, οι μεγάλες αλυσίδες που αναθέτουν σε άλλες εταιρείες να κατασκευάσουν ή να συσκευάσουν. Συνήθως το κάνουν αυτό οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Είχαμε ζητήσει να είναι υποχρεωτική ένδειξη του πραγματικού κατασκευαστή του προϊόντος που δεν είναι η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, είναι κάποιος άλλος που απλώς τα παρασκευάζει για την αλυσίδα αυτή. Αυτά και εδώ δεν καταλαβαίνω τι έχει κάνει η Ευχαριστώ. Κυρία Κλάς.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 να κάνουμε βήματα ο ένας στην κατεύθυνση του άλλου. Δύο-τρία θέματα που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Επιτρέψτε μου να σας πω ποια είναι. Το ένα είναι η σήμανση της ε, προέλευσης. Εγώ προέρχομαι από τη Γεωργία. Εκεί στην περιοχή Άιφελ έχουμε ένα μεγάλο γαλακτοκομείο ε, που μαζεύει γάλα από το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και πού θα γράψει προέλευση. Συλλέγει το γάλα και κάνει ε, το προϊόν. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αρχίσουμε τώρα τα θέματα της περιφέρειας να αναγράφονται από ποια περιφέρεια και από ποια χώρα δεν γίνεται για αυτό το προϊόν. Και έχουμε και ένα τεράστιο πλεονέκτημα διαφήμισης ε, για τις επιχειρήσεις ως Ευρώπη. Αν ε, ο καταναλωτής θέλει οπωσδήποτε να μάθει από πού είναι το προϊόν, μπορεί να το κάνει. Επίσης μπορεί να αγοράζει προϊόντα στο αγρόκτημα, στη λαϊκή, ε, περιφερειακά, επιτόπου. Ας πούμε για το κέτσαπ που είπατε, επειδή δεν γράφει από πού φέραμε τη ντομάτα, αν είναι από τη Χιλή, από την Ισπανία, ε, τότε δεν θα αγοράσω κέτσαπ αν θέλω οπωσδήποτε να γράφει από πού το φέρανε. Ε, η βιομηχανία τροφίμων έχει μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και διαφημιστικό πλεονέκτημα εάν ε, αναγράφει την προέλευση και ακόμα και όταν είναι εθελοντικό δηλαδή και θα θέλει να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Παρακαλώ λίγο να υποχωρήσουν οι συνάδελφοι και να μην το κάνουν πια και σημείο που θα ανατραπεί ολόκληρη η έκθεση κομβικό στην ψηφοφορία. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι οι απομιμήσεις τα υποκατάστατα να αναγράφονται ρητά, ότι, ότι είναι απομίμηση. Και λέει η Ρενάτε Ζώμα ότι έχουν ε, και φαντασία ότι θα γράφει καινοτόμο προϊόν νεωτερικό, μα το προϊόν μαϊμού είναι τελείως διαφορετικό από το ε, καινοτόμο και νεωτερικό. Εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ε, γράφετε τι είναι. Ερζάτς, υποκατάστατο, ξέρω εγώ, τυριού ή προϊόντος. Μετά τον πόλεμο, πριν από πάρα πολλά χρόνια ευτυχώς, είχαμε Ερζάτς καφέ, γιατί δεν είχαμε καφέ και χώριο, ξέρω εγώ, ένα ψεύτικο καφέ. Το ήξερε ο κόσμος ότι δεν ήταν καφές. Λοιπόν, υποκατάστατο ε, τυρού καταλαβαίνει όλος ότι δεν είναι τυρί. Ούτε θα τσακωθώ αν θα μπει στην προστινή στην πίσω πλευρά. Το είπε και η συνάδελφος Χιούπνερ να είναι ευανάγνωστο και θα το βρει ο καταναλωτής. Το παίρνει και στο χέρι του από το ράφι, το κοιτάει και στο μεταξύ ξέρουν οι καταναλωτέ ότι και σημαντικά πράγματα μπορεί να είναι γραμμένα με μικρά γράμματα, αλλά είναι σημαντικά. Και εντάξει, μπορεί ο καταναλωτή να το γυρίσει, εν πάση περιπτώσει, να το δει στην οπίστια πλευρά το προϊόν. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Uh, η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι αναγνωρίζω την εργασία της κυρίας Σόμερ, διότι με μια τόσο περίπλοκη έκθεση δεν είναι καθόλου εύκολο. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Θέλω μόνο να πω πάρα πολύ γρήγορα ότι θέλω να δώσω κι εγώ μερικές προτάσεις, μερικές για την ετικέτα. Αυτό που έχει σημασία είναι η εσωτερική ενιαία αγορά. Δεν μπορούμε να έχουμε τώρα εθνικά πρότυπα που είναι ει βάρο τη εσωτερική αγορά, τη ενιαία αγορά. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και για τι πιο μεγάλε και για του καταναλωτέ. Η ετικέτα λοιπόν, πώ θα είναι αυτή, να είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα του καταναλωτή σε ενημέρωση, χωρί να επιβαρύνεται πάρα πολύ όμω και γραφειοκρατικά και φυσικά Φυσικά η η ετικέτα, γιατί υπάρχει και όριο σε μια ετικέτα και τα πληρώνουν και οι καταναλωτές όλα αυτά, ξέρετε. Το μέγεθος των χαρακτήρων, ε, να είναι ευανάγνωστο. Και εξαρτάται και από τη συσκευασία. Άλλο είναι η συσκευασία 100 ml και άλλο 1 λίτρο. Και πού βάζουμε την προέλευση. Όλο και πιο σημαντική είναι η προέλευση για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα για νοπά προϊόντα, για ψάρια, ε, αλλά και πολλά συσκευασμένα. Βεβαίως να είναι θελοντική αυτή η σήμανση, διότι μπορεί να είναι προστιθέμενη αξία, μπορεί να ενδιαφέρεται η επιχείρηση ακριβώς να αναγράφεται η προέλευση και θα το βάλει αν την ενδιαφέρει την εταιρεία, ακόμα και αν είναι θελοντικό. Από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού στην Ένωση, ε, η ρύθμιση για τα τρόφιμα είναι τεράστια, είναι σχολαστικότατη και εξαντλητική. Οποιοδήποτε προϊόν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προστιθέμενη αξία. Το ξέρουν αυτό πολλοί κατανάλωτες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι ενημέρωση, διαφήμιση ότι είναι καλύτερα τα προϊόντα μας που έρχονται από την Ευρώπη, από εκείνα που έρχονται από τις τρίτες χώρες, τα οποία έρχονται να ανταγωνιστούν τα δικά μας με πιο χαμηλές προδιαγραφές, ενώ οι δικοί μας παραγωγοί παράγουν πολύ πιο ακριβά. Λοιπόν, οποιαδήποτε ενημέρωση, και ακόμα και θελοντική, είναι ευπρόσδεκτη. Γιατί τον ενδιαφέρει να πουλήσει το προϊόν του, να το κάνει πιο ελκυστικό. Αυτά, τα υπόλοιπα τα είπαν οι άλλοι και με κάλυψαν. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Σαπόσκα. Oh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια. Είναι, έχει κρατήσει αρκετά αυτή η συζήτηση. Είμαι όμως πεπισμένη ότι στόχος των συστάσεων αυτών είναι να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές και να προστατευτεί η υγεία τους. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε μόνο για τους καταναλωτές η βλάβη που υφίστανται οι παρασκευαστές δεν είναι απαραίτητη με την επιβολή υπερβολικών ε, ή υπερβολικά αυστηρών περιορισμών και που δεν έχουν αντίστοιχο αποτέλεσμα στους καταναλωτές. Ένας ε, ανεύθυνος κανονισμός δεν θα ε, είναι επιζήμιος στις μεγάλες επιχειρήσεις στο βαθμό που θα βλάψει τις μικρομεσαίες θέλουμε να γνωρίζουμε, ας πούμε, τον ορισμό της μερίδας. Θεωρώ ότι καταρχήν η ποσότητα της μερίδας αναφέρεται πάντοτε στη συσκευασία. Δεύτερον, η ένδειξη αναμερίδα βοηθά τον καταναλωτή να επιλέξει την σωστή τροφή. Τρίτον, αν υπάρχει μόνο ένδειξη για 100, γραμμάρια ή 100 ml, περιπλέκει αυτό και παραπλανεί. Διότι ανάλογα πολύ συχνά η, η ποσότητα που καταναλώνει κανείς είναι πολύ μικρότερη από 100 γραμμάρια ας πούμε μιας τσίχλας. Και τέλος, οι πληροφορίες για τα 100 ml ή τα 100 γραμμάρια που αναφέρονται υποχρεωτικά αναφέρονται ε, στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Άρα ο για τον καταναλωτή η σύγκριση πάντοτε μπορεί να γίνει. Α, και κάτι άλλο. Προσπάθησα να προτείνω στην τροπολογία μου την 302 μια ε, συμβιβαστική λύση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, θα είμαι και εγώ σύντομη. Γιατί ούτω ή άλλω ε, από δύο τελικέ φράσει ε, η αλλω πω δυο αυτή ήταν πολύ μακριά και είδαμε πολλές διαφορετικές απόψεις στην αναζήτηση μιας λύσεις σε προβλήματα που είναι κάποιες φορές πολύ περίπλοκα. Πιστεύω πως ε, η γνώμονάς μας θα πρέπει να είναι το συμφέρον του καταναλωτή καταρχήν. Κάτι που ήδη είναι αρκετά δύσκολο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο private label, κάτι το οποίο ήδη συζητήθηκε, γιατί πιστεύω ότι αυτό που έγινε, που πέρασε μάλλον σε πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, τελικά αφέθηκε κατά μέρο. Ενώ αντίθετα πιστεύω πω είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρον τον καταναλωτή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανεί πέρα από το σήμα του ε, διανομέα ποιο είναι ο πραγματικός ε, διανομεύση. Και επίση είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να γνωρίζει πω ο παραγωγό έχει αλλάξει όταν έχει αλλάξει και άρα να μπορεί να διαπιστώσει την αλλαγή για την ημερομηνία κατάψυξης. Εδώ έχω πρόβλημα γιατί πιστεύω πως μπορεί κάτι τέτοιο να καταστεί διακριτική μεταχείριση σε σχέση με άλλες μέθοδους συντήρησης για τις οποίες δεν ζητείται αυτό το στοιχείο. Επιπλέον γνωρίζουμε πως η κατάψυξη είναι μια τεχνική από τις πιο αποτελεσματικές για να διατηρηθούν οι ιδιότητες των τροφίμων και άρα είναι άσκοπο να επιβαρύνουμε με περαιτέρω κόστος μια τροφική αλυσίδα η οποία προσφέρει πολλές εγγύσεις κυρίως αν τεθούν σε εφαρμογή οι έλεγχοι οι οποίοι προβλέπονται και οι οποίοι είναι απαραίτητοι και σημαντική. Δεν, έχει νόημα να βάζει κανείς μια ημερομηνία που θα μπορούσε, μάλιστα γιατί ξέρουμε πως πολλές φορές η ημερομηνία κατάπτυξης μπορεί να είναι πολύ μακρινή από την ε, πραγματική τοποθέτηση στην ε, πώληση και θα μπορούσαν να προσφέρουν στον καταναλωτή μια μορφή συντήρησης που είναι πολύ καλύτερη από ένα σωρό άλλα είδη συντήρησης όπως ας πούμε τα διάφορα συντηρητικά τα οποία δεν είναι τόσο υγιεινά. Τώρα, ο ευανάγνωστος χαρακτήρας ε, είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ευανάγνωστες οι πληροφορίες. Δεν αρκεί να βγάζει κανείς μια νομοθεσία, δεν αρκεί να μιλάμε μόνο για το μέγεθος των γραμμάτων. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα και έχουμε βρει μια συμβιβαστική με ε, το Συμβούλιο. Υπάρχει ένα τελευταίο πράγμα, ένα τελευταίο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό σημαντικό για μένα και το οποίο πιστεύω είναι λίγο ε, προβληματικό. Το αυτό που λέτε για τη μερίδα ή τα 100 γραμμάρια. Είναι προφανές ότι χρειάζονται τα 100 γραμμάρια για να μπορεί κανείς να κάνει σύγκριση ανάμεσα στα διάφορα προϊόντα. Να μπορεί να δει από τα διάφορα προϊόντα ποια είναι τα ε, στοιχεία. Καλό είναι να ξέρει όμως κανείς και ποια είναι η μερίδα, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα στα μεταπημένα προϊόντα ήδη υπάρχουν μέσα οι, οι μερίδες. Αν έχω ας πούμε κρακεράκια πρέπει, μπορεί να φάω ένα πακέτο και πρέπει να ξέρω πόσα θερμίδες θα πάρω. Αν φάω ένα σοκολατάκι πρέπει να ξέρω πόσες θερμίδες θα πάρω από αυτό το σοκολατάκι. Γιατί δεν πρέπει να πάρω το κομπιουτεράκι και να αρχίσω να κάνω υπολογισμούς πέρα από στην ε, συσκευασία των ε, ε, ζυμαρικών που εκεί τα ζυγίζω γιατί κάνω 100 γραμμάρια το κεφάλι. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, αφού υπάρχουν και μελέτες που έχουν γίνει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενημέρωσης για τα Τρόφιμα, δείχνουν οι μελέτες αυτές πως οι καταναλωτές θεωρούν πως είναι πολύ πιο κατανοητή η πληροφόρηση ανά μερίδα. Πολύ πιο χρήσιμη από ότι η πληροφόρηση για τα 100 γραμμάρια. Μιλάμε λοιπόν για κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Είναι σωστό για τα 100 γραμμάρια, να τα έχουμε και αυτά, αλλά είναι επίση σωστό και πιο ενδεικτικό για αυτό που πραγματικά εισάγουμε, μάλλον ε, ε, ε, καταναλώνουμε, πολλές φορές η μερίδα είναι ειδική. Ε, τρώω τέσσερα μπισκότα το πρωί, ας πούμε, μα δεν παίρνει κανείς ζυγαριά να μετράει και να ζυγίζει τα μπισκότα πρωί πρωί. δεν ξέρω, μπορεί να είναι άλλες συνήθειες σε άλλες χώρες. Ε, κανείς έχει εκεί τη ζυγαριά, ίσως εσείς ε, βγάζετε τα κρακεράκια <laughs> από το πακέτο, τα ζυγίζετε και λέτε «Α, όχι, θα αφήσω δύο κρακεράκια στην άκρη γιατί είναι πιο πολλά από 100 γραμμάρια». Όχι. Ε, οι περισσότεροι παίρνουν ε, την μερίδα όπως είναι ήδη χωρισμένη, προσυσκευασμένη και την καταναλώνουν. Ευχαριστώ. Έφτασα λίγο καθυστερημένα και έχασα ένα κομμάτι της συζήτηση, αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με βάση τα όσα είπε η συνάδελφος Βίλμοντ, γιατί υπήρξαν διάφορες τροπολογίες, ειδικά όσον αφορά την ονομασία προέλευσης, την ένδειξη προέλευσης και η πρόταση του Κοινοβουλίου είναι καλύτερη από αυτή του Συμβουλίου. Και είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε που σφάζεται το ζώο για να είμαστε βέβαιοι πως αποφεύγονται οι, μακρές, ε, οι μακρινές μάλλον μεταφορές. Η Κομισιόν δεν πρέπει τώρα να αρνηθεί την βελτίωση αυτών των κανόνων, γιατί ούτως ή άλλως υποσχέθηκε να προχωρήσει στην βελτίωση. Όσον αφορά τώρα την... Ε, την... και το θεσία, νομίζω πως πολλοί καταναλωτές στην Ευρώπη συμφωνούν και δεν ξέρουν ακριβώς πόσες θερμίδες ε, παίρνουν με τα εινοπνευματώδη ποτά, το αλκοόλ. Σκέφτεται κανείς ας πούμε το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι πολύ πιο υψηλό ε, και όσον αφορά το κρασί και εκείνο έχει πολύ πιο μεγάλη θερμιδική περιεκτικότητα ε, καθώς και η μπύρα ενώ έχουν χαμηλότερο ποσοστό αλκοόλ. Και έπειτα όπως είπε η κυρία Γουίλμοντ και εμείς υποβάλαμε τροπολογίες. Για παράδειγμα στην 152 θέλουμε να στηρίξουμε το γεγονός ότι στο πακέτο στη συσκευασία δεν θα πρέπει να δίνονται παραπλανητικές ε, πληροφορίες. Για παράδειγμα, στην χώρα μου υπάρχουν γλυκά που λέει ότι περιέχουν διάφορους καρπούς, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν οι καρποί. Στη χώρα μου λοιπόν θεωρούμε πως αυτό εντάξει είναι, δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν ε, καρποί μέσα στο γλύκισμα, οι αρχές μας λένε ότι το δέχονται. Η τροπολογία λοιπόν 152 ορίζει αυτά τα οποία εγκρίθηκαν στην πρώτη ανάγνωση. Τώρα για τα vegetarian, τα χορτοφαγητά, έπειτα έγινε λόγος για τα αυγά. Ε, υπήρξε μια πρόταση στην πρώτη ανάγνωση, μα όμως δεν έχει νόημα να υπάρχουν τέτοιες απαγορεύσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Απλά χρειάζεται να γνωρίζει κανείς και να γνωστοποιεί στους καταναλωτές από πού προέρχονται αυτά τα αυγά για να μπορούν να αποφεύγουν ας πούμε, να αγοράζουν προϊόντα με εισαγόμενα αυγά. Αυτά για την ώρα. Κύριος Μαθιουδάκης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούσα αυτή τη συζήτηση. Εν μέρη, συμμερίζομαι την άποψη της κυρίας Ροτμπέρεντ ότι και πάλι εδώ έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατόν να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Προφανώς η Κομισιόν θα το προσπαθήσει αυτό με κάθε τρόπο. Θεωρώ ότι προέκυψαν κάποια ζητήματα ως θεμελιώδους σημασίας, θέματα που κυρίως ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των μελών. Το θέμα καταρχήν της ε, επισήμανσης στο μπροστινό μέρος της συσκευασία. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν είχε στηρίξει την αρχική τροπολογία μάλλον την τροπολογία του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση για μια υποχρεωτική ε, σήμανση στο μπροστινό μέρος της κεμβασίας... για πέντε στοιχεία. Απογοητευτήκαμε μάλλον από το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν συμφώνησε με την πρόταση της Κομισιόν που στήριζε το Κοινοβούλιο, είπαμε ότι θα στηρίξουμε οποιαδήποτε θέση προέρθει επ' αυτού από το Κοινοβούλιο. Επιμένουμε λοιπόν σε αυτό όσον αφορά την σήμανση στο μπρος μέρος της συσκευασία. Τώρα, όσον αφορά την χώρα προέλευσης, εδώ είναι προφανής μια διάσταση απόψεων. Τα επιχειρήματα κάθε πλευράς κατανοητά. Πολλοί καταναλωτές ζητούν να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια Αυτό είναι πολύ δύσκολο και για τους παραγωγούς και για τους παρασκευαστές των προϊόντων. Αυτό που προέκυψε από το Συμβούλιο θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Και αυτή η θέση θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Κοινοβούλιο να θεωρηθεί μια συμβιβαστική λύση. Τώρα, το ευανάγνωστο. Χαιρόμαστε που αναγνωρίζετε αυτό το θέμα. Επίσης χαιρόμαστε που διαπιστώνουμε ότι η η συγγήτρια ε, προτείνει στήριξη της θέσεως του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Αυτά θεωρούμε τα σημαντικότερα στοιχεία της συζήτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει πάλι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε ότι παρότι το έχουμε συζητήσει πολύ, χρειάζεται ακόμα συζήτηση το θέμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω καταρχάς αυτό που είπε η Κρίστα Κλάς. Είναι δεύτερη ανάγνωση τώρα. Και στη δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να σκέφτονται όλοι τι ε, πνεύμα συμβιβασμού θα επιδεικνύουν. Δεν μπορεί να κάνει πάντα ο ένας βήματα στην πλευρά του άλλου, θα πρέπει και ο άλλος να δείξει μια προθυμία, έτσι δεν είναι. Και ελπίζω αύριο με τους σκιώδεις ηγητές της συνεδρίαση που θα έχουμε να καταφέρουμε να ε, κάνουμε βήματα ο ένας προς τον άλλον, να τα βρούμε κάπου. Χρονολογικά, με τη σειρά δηλαδή που μίλησαν οι συνάδελφοι, θα απαντήσω. Η Γκλένις Βίλμοτ μίλησε για τα τρανς λιπαρά ότι θα πρέπει να αναγράφονται, συμφωνώ και επιμένω κι εγώ σε αυτό, αλλά ε, για μένα δεν έχω μεγάλη σημασία, δεν έχω ιδιαίτερη άποψη, αλλά είναι λέει και τεχνικό το πρόβλημα. Είναι τα τεχνητά τρανς λιπαρά και τα φυσικά. Τα φυσικά από τα λιπαρά δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε και υπάρχουν πολλά προϊόντα, το είπε και ένας συνάδελφος προηγουμένως, που περιέχουν τρανς λιπαρά από τη φύση τους. Και αν αναγράφεται, αυτό είναι γάλα και γαλακτοκομικά. Αυτό θέλουμε να αναγράφεται και να έχουμε αρνητική εικόνα στους καταναλωτές ότι περιέχει τρανς λιπαρά, αφού είναι φυσική η παρουσία τους και δεν αποφεύγεται και στο γάλα και στα γαλακτικομικά. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Υπάρχουν τεχνητά, τρανς λιπαρά και φυσικά, αλλά δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Ποιο είναι φυσικής προέλευσης και ποιο είναι. Και λογικά και μόνο. Πώς να απαγορευτεί αυτό. Ε, το θεωρώ ανεδαφικό. Δεν μπορούμε να τις απαγορεύσουμε αυτές τις ουσίες, αφού είναι από τη φύση τους σε μερικά προϊόντα. Ε, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και περαιτέρω, θέλετε. Δεν με πειράζει αυτό, δεν θα μας ε, οδηγήσει αυτό στη συνδιαλλαγή. Για την πληθώρα των τροπολογιών, όντως, ως εισηγήτρια, κατέθεσα και εγώ πολλές δικές μου τροπολογίες. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ε, το Συμβούλιο Υπουργών μέλησε πάρα πολλές λεπτομέρειες και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι ε, πανυπέβαλαν τροπολογίες από την πρώτη ανάγνωση και καλώ έπραξαν. Σωστό είναι και αυτό. Το είχαμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν. Και ε, αντιπαρατηθήκαμε κιόλα. Θα ήθελα να πω ότι εκτός από την έκθεσή μου έχω κάνει περίπου 30 επιπλέον τροπολογίες που είναι αμυγός τεχνικής φύσεως. Παρακαλώ να το λάβουν υπόψη οι σκιώδες ηγητές. Πρόκειται και πάλι για προσαρμογές στις καινοτομίες που έχει επιφέρει η ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Η νομική υπηρεσία μου υπέδειξε ότι χρειάζονται αυτές οι τεχνικές προσαρμογές. Να αλλάξω έτσι τις τροπολογίες λόγω της συνθήκης Λισαβόνας. Παρακαλώ, σκεφτείτε αυτό, δεν αλλάζει το περιεχόμενο. Είναι αμυγός τεχνική προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, ε, η επισήμανση Τη πρόελευση. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτό και μάλιστα είπαν ότι είναι σημαντικό για τον καταναλωτή. Το ακούω εγώ από διάφορε συζητήσει, το συζητάω με πάρα πολλού και το ξέρω κιόλα ότι είναι σωστό. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε εάν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι σημαντικό για όλους τους καταναλωτές. Είναι πολύ λίγες οι μελέτες που έχουν γίνει, σε λίγα κράτη-μέλη επίσης και για το θέμα ε, προέλευση, σήμανση είναι σημαντική αυτή για τον καταναλωτή και διαπιστώθηκε μάλλον ότι για τον καταναλωτή είναι ασήμαντο από τις έρευνες φάνηκε. Τώρα εξαρτάται σε ποιες χώρες έγινε αυτή η έρευνα και από ό,τι φαίνεται και το πιστεύω αυτό που λένε οι συνάδελφοι, σε ορισμένες χώρες Καταναλωτέ νοιάζονται πολύ περισσότερο για την προέλευση και σε κάποιες άλλες λιγότερο. Στη Γερμανία οι περισσότεροι καταναλωτέ, η μάζα, δεν ενδιαφέρεται για την προέλευση του προϊόντος, ενδιαφέρεται για την τιμή του προϊόντος. Το πορτοφόλι μετράει και η τσέπη. Σε άλλες χώρες, αν ισχύει αυτό, το δέχομαι, αλλά ε, δεν έχουμε ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση αυτό. Είναι προσωπική παραδοχή πολλών και Πολλές ε, οργανώσεις ε, προστασίας των καταναλωτών ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, ε, μας τα διηγούνται αυτά, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Ο κύριος Μαθιουδάκης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής σωστά είπε, ξανά όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι η αναγραφή της προέλευσης μπορεί να έχει και το εξής πρόβλημα γραφειοκρατία και φόρτος υπερβολικός. Αυτό είναι πρόβλημα σίγουρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι ο τομέας των τροφίμων σε ποσοστό 80% απαρτίζεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε θα πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Και τελικά, και να έχουμε πάντα υπόψη μας, όλα τα πληρώνει ο καταναλωτής τα επιπλέον για μια επιπλέον σήμανση με πούμε, τη χώρας προέλευσης. Δεν το πληρώνουν οι οι εταιρείε, μετακυλίουν το κόστος. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας πάντα. Αλλά φροντίσουμε, όπως είπαμε, να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Επειδή τη αρχή δεν διαφωνώ. Και πρέπει να το ξαναπώ εδώ. Ε, προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να είναι εφικτό αυτό. Και να είναι και σε ένα λογικό κόστος. Έτσι χρειάζεται και άλλη συζήτηση και αυτό ενδεχομένω και με το Συμβούλιο Υπουργών. Για το μέγεθος της μερίδας τώρα υπάρχει μια πρόταση, δική μου αρχική έτσι κι αλλιώς, να ορίσουμε ποια είναι η θερμίδα, πόσο είναι μια, μια μερίδα, συγγνώμη. Μπορεί κανείς να, ότι είναι η φέτα, το φλιτζάνι, το κουταλάκι του γλυκού ή το κουταλάκι της σούπας. Η φέτα όμως ε, μπορεί να είναι μερίδα εφόσον το προϊόν κυκλοφορεί σε φέτες. Γιατί άμα αγοράσω ένα τυρί ή ένα ψωμί, το μέγεθος της φέτας το καθορίζω εγώ. Και επίσης το κουταλάκι του τσαγιού, του καφέ και το κουτάλι της σούπας επίσης δεν είναι ενιαίο μέγεθος σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό είναι πρόβλημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει και αυτό, ότι η μερίδα είναι μια μερίδα που μπορεί να φανταστεί ο καταναλωτής. Άμα το βάλουμε σε γραμμάρια, ο καταναλωτής δεν έχει στο μυαλό του πόσο είναι γραμμάριο. 25 γραμμάρια πόσο είναι δηλαδή. Ε, είναι ένα πιάτο ε, βαθύ, γεμάτο. Είναι μια παιδική χούφτα γεμάτη. Πρέπει τη μερίδα να την ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους με όλους τους ενεχομένους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται αυτό και μετά να δουλέψουμε με βάση τη μερίδα. Από την αρχή είπα ότι είμαι πρόθυμη να αναγράφεται αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά να το ορίσουμε. Αλλά να μην ωρεοποιούνται ε, με πολύ μικρές ε, μερίδες για τη συγκρισιμότητα οπωσδήποτε να γράφεται ένα 100 γραμμάρια η θρεπτική αξία, η θερμιδική αξία. Το αποφασίσαμε αυτό. Το προτείνει άλλωστε και το Συμβούλιο. Και στον πίνακα της θρεπτικής αξίας υποχρεωτικά ε, στο πίστιο μέρος της συσκευασία. όπου σκεφτόμαστε να βάλουμε και τη μερίδα. Ξέρετε ότι έχει γίνει ένα λόμπι και συνεχίζεται αυτό το καιρό μαζικά πίεση στην πρόστια πλευρά να μην αναγράφεται μόνο αυτό το θέμα του, των 100 γραμμαρίων, αλλά και ε, μερίδες. Αλλιώς ε, κατηγορούνται, λέει, ορισμένα προϊόντα ε, επειδή έχουν πολλές θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Όλα αυτά που συζητάμε είναι για το πρόστιο μέρος της συσκευασίας Στο πίσω θα μπει έτσι κι για τα χρωστικά τρόφιμα. Το είχα συζητήσει και εγώ με τις ε, τροπολογίες αυτές, με τους συντάκτες δηλαδή. Χρειάζεται διευκρίνηση, το έχω γράψει και στη λίστα μου για τα θέματα που θέλω να συζητήσω με τους σκιώδες αύριο. Χρειάζεται διευκρίνηση. Στη σημερινή συνεδρίαση πήραμε αυτό το χαρτί από μια συμμαχία για τη διαφάνεια στα τρόφιμα σαν μη κυβερνητική οργάνωση ακούγεται, που δεν είναι και το θεωρώ και εγώ αισχρό. Ε, είναι απαράδεκτο είδος άσκησης πίεσης αυτό. Και επίσης δεν θεωρώ σωστό να μας μοιράζουν οι συνάδελφοι χαρτιά στα έδρανά μας, γιατί το είδαμε και αυτό στην πρώτη ανάγνωση και αυτό με ενοχλεί. Λοιπόν, για τα τρόφιμα που είναι χρωστικές ουσίες και πάλι είναι εδώ αντικρούωμενα τα συμφέροντα στη βιομηχανία όπως καταλαβαίνετε και έχω λίγο ένα πρόβλημα εγώ αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε και αύριο με τους σκιώδες ηγητές, ότι και αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό. Όταν διαφημίζω, ας πούμε, ότι οι χρωστικές μου είναι μόνο φυτικής προέλευσης και έχω ένα ωραίο χρώμα στο προϊόν, αυτό μπορεί να δείχνει ότι έχει μέσα ε, πολλά κομμάτια φρούτο και να μην είναι έτσι. Και το άρθρο 7 στον κανονισμό Τώρα, για το ευανάγνωστο, το μέγεθος των χαρακτήρων των γραμμάτων, θέλουμε να είναι ευανάγνωστο και όχι μόνο το μέγεθος ε, της γραμματοσυράς, αλλά να υπάρχει και ένα κοντράστ, μία αντίθεση οπτική ε, ανάμεσα ε, στη γραφή, τη γραμματοσυρά και το φόντο για να είναι ευανάγνωστο. Βεβαίως, ο συμβιβασμός έχει πολλά στοιχεία, εκτός από το ευανάγνωστο, η απόσταση των γραμμάτων, το ένα από το άλλο, ή των αριθμών, του ενός από, το, από τον άλλον αριθμό. Η Ευρωπαϊκή τον αλλον αριθμο μιλάει για δεσμευτικούς κανόνες, binding rules. Και τους εκπονεί κιόλας για το τι είναι ευανάγνωστο. Και αυτός είναι ο σωστός δρόμος, ο καλύτερος πιστεύω το μέγεθος των χιλιοστών, το μέγεθος των χαρακτήρων είναι τόσο τεχνικό ζήτημα που ως κοινοβούλιο δεν είμαστε σε θέση να το αποφασίσουμε. Αυτό είναι θέμα ειδικών. Συνέβη και αυτό και ε, γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση του Συμβουλίου και αυτό είναι και ε, κάτι που αφορά και το μέγεθος της συσκευασίας. Για πολύ μικρές συσκευασίες προτείνονται και μικρότεροι χαρακτήρες και οι πάρα πολύ μικρές να εξαιρούνται από τις διάφορες διατάξεις, γιατί δεν χωράει όλο αυτό που θέλουμε να γράψουμε στη συσκευασία. Κατά τα δεν νομίζω να απέχουμε πάρα πολύ στις απόψεις μας εδώ. Θέλω να πω στην κυρία Γκροστέτ ότι η σήμανση ειδικών τροφίμων, ας πούμε για βρέφη, είναι σε άλλη νομοθεσία ρυθμισμένο. Και εδώ ε, αυτό δεν θα πρέπει να το θίξουμε είναι προφανές και αυτονόητο και ούτε θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα. Η ε, συνάδελφος ε, Γροστέτ μίλησε και για το νάτριο. Να αναφέρεται επιπλέον η συγκέντρωση του ή η περιεκτικότητα του τροφίμου σε νάτριο. Από πλευράς επιστημονικής είναι σωστό να αναφέρουμε τη συγκέντρωση νατρίου, όχι το αλάτι. Αλλά εμεί είπαμε να γράφουμε αλάτι γιατί ο καταναλωτής το καταλαβαίνει καλύτερα. Τώρα πόσο νάτριο έχει και πόσο από φυσικέ πηγές, ξέρω εγώ γιατί και αυτό ακούγεται. ενημερώνει και για την ίδια τη φύση του προϊόντος, αλλά και για άλλες πηγές νατρίου, πλην του άλατος. Το αλάτι έχει νάτριο 40%, αλλά υπάρχουν και άλλες πηγές νατρίου άλλες ενώσεις του ο, νατρίου, γλουταμάτ, ξέρω εγώ και τέτοιου τύπου ενώσεις. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί πάρα πολύ, όμως θα τα δούμε και εκεί αυτά. Για την εσωτερική αγορά είπατε ότι θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Το είπε ο κύριος Κράμερ και εγώ συμφωνώ, με ενδιαφέρει και εμένα πολύ αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να πάρουμε τις αποστάσεις μας από αυτό που ακούγεται ε, τα κράτη να έχουν τη δυνατότητα να βάζουν ε, σούπερ ε, δικές τους ρυθμίσεις επιπλέον. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιβαρυντικό. Μα τα είχαμε πει αυτά και στην πρώτη ανάγνωση και το είχαμε απορρίψει σε μεγάλο βαθμό. Τι άλλο έχουμε. Ο κύριος Ρώση μίλησε για τα duty free για τα αφορολόγητα προϊόντα. Äh, äh, Να. Είναι μόνο στα αγγλικά τα αφορολόγητα είδη που πολλούνται μόνο στα αεροδρόμια και εκεί που πολλούνται αφορολόγητα είδη. Να είναι μόνο στα αγγλικά. Θα το συζητήσουμε αυτό. Ναι, έχει νόημα σε μεγάλα διεθνή αεροδρόμια. Όχι μόνο στη γλώσσα της χώρας αλλά μπορούμε και από αυτού να συμφωνήσουμε και να πούμε τη γλώσσα της χώρας είναι αγγλικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά θα ήταν νόημα να επιμείνουμε να είναι μόνο στη γλώσσα της ε, λόγω χώρας. Α, για το κινηματογράφο Multiplex, το είπε ο συνάδελφο Κυλακάκη, ο οποίο έχει φύγει στο μεταξύ. Εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση ω αιτιολογική σκέψη. Εντάξει. Και τώρα ξανάρχεται να ψηφιστεί. Θέλω ξαναπώ στο συνάδελφο Ρώση. Οι ημερήσιες ανάγκες μιας ενήλικης γυναίκας. Ελπίζω να σας κατάλαβα καλά. Διαμαρτύρεστε ότι μόνο, μιλάμε μόνο για τη γυναίκα. 2.000 θερμίδες θα πρέπει να υπάρχει για τον άνδρα ξεχωριστή αναφορά. Αλλά η προτινόμενη μερίσια ε, ανάγκη ε, αναφέρεται σε γυναίκες. Αυτό είναι το μέγεθος. Γι' αυτό πρέπει να το γράφουμε. Και ο καθένας προσωπικά ε, μπορεί να διαφέρει στην ημερήσια προτινόμενη κατανάλωση. Ας πούμε, ε, έχουν άλλες ανάγκες από ό,τι οι γυναίκες και μάλιστα ανάλογα και με την ηλικία διαφέρουν. για την ημερομηνία λήξεως. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα με προϊόντα που έχουν πολλά συστατικά ή διαφορετικά συστατικά. Και αυτό το συζητούμε και θα χρειαστεί διευκρίνηση. Είναι γνωστό, έχει αναγνωριστεί το πρόβλημα. Η ημερομηνία ψήξης ή κατάψυξης είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κρέας μόνο. Γι' αυτό κατατέθηκε αυτή η τροπολογία, έτσι δεν είναι, και μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό. Μετά ρώτησε ο συνάδελφος Ρώση, τι γίνεται με νοπά προσυσκευασμένα τρόφιμα, τι είναι αυτό. Το λέει μια τροπολογία μου αυτό. Εξαιρούνται τα προϊόντα που κυκλοφορούν χήμα. Αλλά υπάρχουν προϊόντα που συσκευάζονται εκείνη την ώρα για να αγοραστούν στα σούπερ μάρκετ. Ας πούμε ε, διάφορες σαλάτες που παρασκευάζονται και τις πουλάνε σε πολύ μικρές συσκευασίες για την ίδια κατανάλωση της ημέρας. Μετά, η μάρκα του παραγωγού, του παρασκευαστή, η ίδια μάρκα. Ας, ξέρουμε στα σούπερ μάρκετ ότι έχουν δική τους ετικέτα, η, ε, ίδια ετικέτα της εταιρεία και πάλι είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα. Πάρα πολλοί ε, παραγωγοί λένε ότι δεν θέλουν να μπει το όνομά μας εκεί, η μάρκα μας, γιατί εμείς παράγουμε για διάφορες αλυσίδες ε, σούπερ μάρκετ με διάφορους αποδέκτες ανάλογα με το τι θέλει ο κάθε καταναλωτής. Και επιπλέον δεν θα ήταν καλό για μας να επιμείνουμε ε, πάντα να αναφέρονται ε, τα δικά μας στοιχεία ή το δικό μας όνομα σε φθηνά προϊόντα που πουλάει ε, ένα σούπερ μάρκετ με ίδια ετικέτα. Οπότε ο κόσμος δεν θα αγοράζει το δικό μας γνήσιο προϊόν, αλλά θα αγοράζει το προϊόν του σούπερ μάρκετ με την ονομασία του σούπερ μάρκετ και το δικό μας όνομα. Γιατί το δικό μας είναι πιο ακριβό με τη γνήσια ε, ονομασία και ετικέτα. Και από αυτό βγάζουμε λιγότερα χρήματα. Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Και ένα τελευταίο. Πρότεινε Κρίστα να γράψουμε υποκατάστατο τυριού. Δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη τυρί για ένα προϊόν που δεν είναι τυρί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας πούμε, πώς να το πω Δεν μπορώ ένα σκεύασμα που δεν είναι ζαμπόν να το βαφτίσω ζαμπόν επειδή έχει μορφή ζαμπόν. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση, αλλά ε, δεν γίνεται να φέρει την ονομασία αυτή ένα προϊόν που δεν είναι αυτό το προϊόν. Αυτά νομίζω ήταν τα σημαντικότερα που ε, αναφέρθηκαν και ένα τελευταίο να τονίσω Νομίζω ότι θα πρέπει επιγόντως να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα σε δεύτερη ανάγνωση. Να συμφωνήσουμε δηλαδή και να μην πάμε στη συνδιαλλαγή. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι θετική η έκβαση της συνδιαλλαγής, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι μπορεί να αναβαγίσει και μια συνδιαλλαγή αν είναι τόσο ανένδοτες ε, οι θέσεις. Νομίζω ότι σε δεύτερη ανάγνωση μπορούμε να βρούμε λύσεις συμβαστικές και με το Συμβούλιο. Γιατί αν να βαγίσει η διαλλαγή θα πρέπει ο καταναλωτής να περιμένει άλλα δέκα χρόνια για καλύτερη σήμανση στα τρόφιμα και δεν νομίζω ότι επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε χρόνο. Έλπιζα να μπορέσουμε να κλείσουμε, αλλά κυρία Τέρες ζήτησε το λόγο συντομία. Α, κύριος Τέρες. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ε, όσον αφορά την επισήμανση για τη χώρα προέλευσης. Προέδρευσα στις συνεδρίες του Χονγκ Κόνγκ. το 152 χώρες. Συμφωνήσαμε θα μπορούσε να υπάρχει σήμανση για τη χώρα προέλευσης ακόμα και αν ένα ζαμπόν έχει παραχθεί στο Καναδά. Ε, τι γίνεται έπεσε μια πινακίδα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος, κανένα σούπερ μάρκετ και αυτό δεν θα στοιχίσει παραπάνω, γιατί έχουμε την, στο κρασί τη σήμανση προέλ... χώρα προέλευση. Στο σούπερ μάρκετ, α πούμε, λέμε γαλλικό, ιταλικό κτλ. Δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ε, Σαφώ στο Χονγκ και παρά την αποτυχία τη Ντόχα, Είναι δεν υπάρχει πρόβλημα με την επισήμανση για τη χώρα προέλευσης. Ωραία. Τώρα θα ψηφίσουμε. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 19. Είχα πει ότι δεν θα ξαναρχίσουμε καινούργια συζήτηση. Ε, θα ξαναμπεί στην μέρη σε διάταξη. Η για να πει κάτι άλλο. Ε, Ο συνάδελφος Στέρντι δεν είναι τόσο δύσκολο σε νοπά προϊόντα και σε χήμα προϊόντα θέλετε, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι τα επεξεργασμένα προϊόντα, τα μεταποιημένα προϊόντα, που είναι άλλη ιστορία, γιατί έχουν διάφορα συστατικά και ορισμένοι θέλουν να ε, αναγράφεται η πρόληψη του κρέατος, άλλοι λένε του κυρίου, του βασικού συστατικού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Το είπαν πολύ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τα άλλα, αλλά θα το ξανασυζητήσουμε, δεν τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στις 19 Απριλίου στην Ολομέλεια θα εισαχθεί τον Ιούλιο το θέμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Είναι η εκτελεστική πράξη για ζωοτροφές και τρόφιμα από την ε, Ιαπωνία μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα. Ο κύριος Φλου από την Κομισιόν έχει καταρχήν τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζετε, στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα είπαμε ότι θα ευθυγραμμίσουμε τα αρχικά μέτρα που ελήφθησαν και που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν στις 25 Μαρτίου για να συνταχθούν με τα μέτρα που έλαβαν οι Ιαπωνικές αρχές μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα. Χτες η Κομισιόν ενέκρινε μια τροπολογία, ένα μέτρο προστατευτικό που εφαρμόζει τα μέτρα που αποφάσισαν οι Ιαπωνικές αρχές για το ιόδιο και για το κέσιο. Αυτό αφορά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που εισάγονται από την Ιαπωνία και που για, αυτά, για αυτές ισχύουν αυτά τα οποία επιβλήθηκαν για την εσωτερική αγορά της Ιαπωνίας. Γιατί τα δικά μας επίπεδα ήταν διαφορετικά από αυτά τα Ιαπωνέζικα. Δηλαδή μπορούσαμε να εισάγουμε προϊόντα που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στην εσωτερική αγορά της Ιαπωνίας. Το νέο αυτό μέτρο δεν αλλάζει τίποτα. όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστοποίησης που έχουμε επιβάλει στην Ιαπωνία, ότι τα προϊόντα προέρχονται από την Ιαπωνία πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από τις Ιαπωνικές αρχές ότι ως μορφούμενα με τα μέτρα που αφορούν ε, την περιολόγος, περιοχή και επίσης ε, δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το σημείο εισόδου όπου απαιτείται δειγματοληπτικός έλεγχος. Τα μέτρα αυτά με την ευθυγράμμιση αυτή που έγινε είναι μέτρα ανάλογα του κινδύνου. Αναγνωρίζεται επίσης ότι από τη ευθύς εξ αρχής η Ιαπωνία ενημέρωσε, ενημέρωνε την Κομισιόν για τα μέτρα που ελάμβανε. Ποτέ δεν επέτρεψαν σε προϊόντα που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ιαπωνική αγορά για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα, πλέον υπάρχει μία συνέπεια ανάμεσα στον έλεγχο πριν από την εξαγωγή που πραγματοποιείται στην Ιαπωνία και στον έλεγχο που πραγματοποιείται στην Ευρώπη. Επίσης, οι Ιάπωνες θα ε, ε, εφαρμόσουν τα επίπεδα σε προσωρινό επίπεδο, αλλά από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Ιαπωνία αυτά τα μέτρα. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ελέγχουν τις εισαγωγές από την Ιαπωνία. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής δείχνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα επίπεδα ήταν είτε μη ανιχνεύσιμα είτε αμεληταία. Ο κύριος Μπαρόζο επίσης ανακοίνωσε ότι τα επίπεδα που καθορίζει ο κανονισμός 3954 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επανεξεταστούν από ειδικούς επιστήμονες στο ερχόμενο διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι όλο και λιγότερα τα παραδείγματα ευτυχώ, αλλά εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν χάσει εντελώς την επαφή τους με την πραγματικότητα. Τελείω όμως. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι έμεινα άναυδη όταν πριν από κάποιες εβδομάδες είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ρύθμιση πριν από 25 χρόνια αυτό που ίσχυε, το έβαλε στο τραπέζι, το έβγαλε από το σιρτάρι, ωραία, ισχύει ακόμα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και τώρα, είπε. Κοιτάξτε να δείτε, περί τίνος πρόκειται. Γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ωριακέ τιμέ και όχι μόνο, αλλά τι λένε οι επιστήμονε ότι είναι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Γνωρίζουμε ότι οι επιστήμονες στην Ευρώπη συμφωνούν. Και αυτό που λέμε ως σύσταση και για την Έύσα στο παρελθόν δεν είναι ε, μονοσήμαντο και αναμφισβήτητο. Είτε είναι αυτό για τα μεταλλαγμένα είτε όχι. Και όταν πρόκειται για επιβάρυνση, ε, μόλυνση τροφίμων με ιόδιο και ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, όπου ο, όλος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, εντάξει, μπορεί να έχει τρομοκρατηθεί και να λέει τι, τι θα κάνω με το ρύζι, τι να κάνω με το πράσινο τσάι, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας σερβίρει τη ρύθμιση για το Τσέρνομπιλ. Δεν λέω ότι είναι καιροσκοπία, αλλά έχω πραγματικά μείνει έκπληκτη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακτήσει την επαφή της με την Ευρώπη, με την πραγματικότητα της Ευρώπης και των βουλευτών. έχει γίνει χαμός τώρα τις τελευταίες εβδομάδες και μας λέτε ότι α, μήπως δεν είναι σωστή εικόνα να έχουμε πολύ χαλαρότερα όρια από ό,τι του Ιάπωνες. Τι ωραία ιδέα. Θα μπορούσα να το είχα σκεφτεί και μόνη μου όμω. Δεν θα έπρεπε να επέμβει ο κύριο Μπαρόσο γιατί το θεωρεί σούπερ ευκαιρία επικοινωνίας. Μα πώ να πάτε να το εξηγήσετε στον πληθυσμό. Είναι τόσο ανεπαρκή αυτή και τόσο μαζεμένη η λιθιότητα, λυπάμαι που το λέω, ε, το λέω σπάνια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα τελευταία χρόνια τα πάμε με λίγα, αλλά αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλη τσαπατσουλιά, είναι πολύ κακή δουλειά και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Συγγνώμη τώρα που τα ακούτε εσείς, κανονικά πρέπει να τα ακούσει ο Επίτροπος, τουλάχιστον, αλλά να τα πείτε και στον κύριο Μπαρόσο ε, που δεν είναι και αιχμή του δόρατος της προστασίας των καταναλωτών, δεν θα τον κατηγορήσει κανείς γι' αυτό, αλλά ε, ακόμα και ο κύριος Μπαρόσο κατάλαβε ότι είναι κακή αυτή η κατάσταση και από πλευράς δημοσίων σχέσεων, ότι κοιτάξτε ακόμα και οι Άπωνες έχουν αυστηρότερα όρια και εμείς όχι. Λοιπόν, να δούμε τι λένε οι επιστήμονες. Ό,τι και να πούν οι επιστήμονες, υπάρχει η αρχή της προφύλαξης. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί επιστήμονε Να του εξηγήσουμε τι είναι αρχή τη προφύλαξη του λέω και στο ΕΨΑ. Τι είναι αυτό λέει το precautionary principle. Να σα πω τι είναι. Φροντίστε πριν ξανάρθετε και μα φέρετε τίποτα στο μέλλον να το έχετε στεφτεί δύο-τρει φορέ και να έχετε συζητήσει και με τις άλλες γενικές διευθύνσεις που καθημερινά έρχονται σε επαφή και με τρόφιμα και με βουλευτές και με εκλογικές περιφέρειες και συνεννοηθείτε λίγο και σκεφτείτε αν ήταν λογικά αυτά που μας φέρετε εδώ. Η κυρία Γκρούστετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να αναφέρω ένα-δύο θέματα δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικά, αλλά το να μιλάμε για τη ρήψη ραδιο, ραδιενεργών ε, αποβλήτων στον ειρηνικό. Μα ε, τα ψάρια είναι αποδημητικά ήδη. Ε, ε ταξιδεύουν, κάνουν και μακριά ταξίδια. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα προσέχουμε μόνο τα ψάρια τα οποία αλλιεύονται στα ιαπωνικά είδωτα, αλλά τι θα γίνει με τη ραδιενέργεια που μπορεί να βρούμε στα ψάρια που αλλιεύονται στα ανοιχτά της Κορέας ή της Κίνας, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν ίσα ίσα χίλια χιλιόμετρα χωρίζουν το βόρεια της ε, Ιαπωνίας από τη Σεούλ. Δεν νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα ειρηνικό. Θα έχουμε πραγματικά όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά την αλληλεία που θα γίνεται στα νερά αυτά, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα ύδατα, όπου μπορεί να βρεθούν όμως τα ψάρια τα οποία αμολύνθηκαν. Αυτά είναι ε, ε, τα ερωτήματα που θέλω να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. undrar kommissionen ο, κύριος Λούτερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να επαναλάβω μόνο το εξής. Αναφέρατε την ε, Ραδινέργεια, μα δεν μπορούμε να πάρουμε κατόφλια 25 ετών, γιατί Πρόκειται για έναν κανονισμό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 25 χρόνια. Ήταν ε, ο κανονισμός Τσερνομπίλ που παγόρεψε τις εισαγωγές από όλες τις τρίτες χώρες. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το ποια κατόφλια θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουν αυξηθεί τα κατόφλια. Πολύ κακή ενημέρωση είναι αυτή. Πρόκειται για παλιά κατόφλια που χρονολογούνται εδώ και 25 χρόνια και αν είχαμε την ίδια πολιτική για το μόλυβδο θα είχαμε πολύ ψηλά κατόφλια για τον μόλυβδο. Τα αλλάξαμε όμως αυτά γιατί είχαμε νέες πληροφορίες επιστημονικές. Και αν κάποιοι απορροφήσουν πολύ ψηλή δόση, αυτό συχνά είναι αντίστοιχο με τις ζημιές σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχουν όμως απορροφήσει χαμηλότερες δόσεις. Αυτό είναι όμως πολιτικό ζήτημα το πώς προσαρμόζει κανείς τα επίποδα κινδύνου και πώς το φορτώνουμε το ανασωπητικό σύστημα πολύ συχνά ένα πολύ με μικρό ποσοστό μόλιβδο ας πούμε στο νοσοποιητικό σύστημα μπορεί να καθορίσει τη διαφορά ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια. Ε, ε, πρέπει δηλαδή κανείς ε, νομίζω να είναι ψύχρεμο. Αντιδράσαμε με γρήγορα στην Ιαπωνία, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να φέρουμε μόνιμε αλλαγέ και ενημερώσει στον κανονισμό. Επίση, διαρωτώ με διότι το κέσιο δεν πρόκειται να εξαφανιστεί μέχρι τον Ιούνιο. Τι κάνουμε λοιπόν για να έχουμε μια πιο μόνιμη λύση για όλα αυτά, μια πιο μόνιμη απάντηση. Φλόρενς, και εγώ συνήθως χαίρομαι πολύ λίγο να κολλάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτή τη φορά δεν έγιναν τα πράγματα όπως παρουσιάστηκαν εδώ. Από τη μια μέρα στην άλλη Ανατράψαν τα πράγματα στην Ιαπωνία ε, και στην Ευρώπη 26 χρόνια δεν χρειαζόμασταν τέτοιους κανόνες. Μετά το Τσέρνομπιλ πήραμε κάποιες ρυθμίσεις σε περίπτωση που γίνει κάτι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν είναι μεγάλη η ακτινοβολία ανεβάσαμε τις οριακές τιμές. Δεν ξέρω αν είναι αυτό καλό ή κακό, δεν το αξιολογώ. Αυτή την έκθεση την έβγαλε από τα συρτάρια της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν σωστό, γιατί αν δεν το είχε κάνει δεν θα υπήρχε καμία ρύθμιση. Αυτό το βήμα ήταν σωστό. Το γεγονός όμως ότι δεν το δούλεψαν τα τελευταία 20 χρόνια μπορεί κανείς να το προσάψει, αλλά θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα και αν ήταν πολύ διαφορετικότερο. Δηλαδή, Ντάκμαρ, εμείς γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Εσύ είσαι και φίλη των Πρασίνων και ο πράσινος Φλόρεντς ε, στη Τζεντεού ε, ήταν ο κακός. Αλλά τώρα δεν είναι η κακή της υπόθεσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πράγμα που δεν θα πρέπει να την εμποδίσει να εργαστεί και εντατικά στο μέλλον. δεν αξίζει, Ντάγμα, να της επιτίθεσε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνήθως συμφωνώ μαζί σου, αλλά σήμερα όχι. volevo Ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη παρέμβασης και εφαρμογής. Των όσων αποκομίσαμε από την εμπειρία του Τσέρνομπιλ και πιο συγκεκριμένα την ανάγκη για ένα πλήρες πλαίσιο όσον αφορά τις ανεκτές δόσεις για τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τους κινδύνους όσον αφορά τις ε, δόσεις στα τρόφιμα. Ιδιαίτερα αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί πολύ είναι η ενδεχόμενη μόλυνση στα κατεργασμένα τρόφιμα και κυρίως αναφέρομαι στο πρόβλημα της ε, κονσερβοποίησης ε, του ψαριού ή του κρέατος που μπορεί να οδηγήσει σε διάδοση ραδιενεργών υλικών και που άρα θα πρέπει να πλαισιωθεί από μια περαιτέρω Ε, διάταξη για τη διαδικασία ε, απορρόφησης της ραδιενέργειας από, τους, ε, από τον ανθρώπινο οργανισμό και άρα να υπάρχει ενημέρωση για τις εσωτερικές δόσεις που μπορεί να οφείλονται στην ε, απορρόφηση αυτών των ραδιενεργών υλικών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όντως μπορεί να αντιμετωπιστεί επί τη βάση της εμπειρίας του Τσινομπίλ, αλλά που προφανώς και εμείς εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι Πιθανότατα βρισκόμαστε ενώπιον ε, μιας ε, νέας κατάστασης γιατί έχουμε προϊόντα σχάσεις τα οποία ίσως είναι διαφορετικά, έχουν διαφορετική συμπεριφορά από το Τσέρνομπιλ. Γι' αυτό και ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν τι σκοπεύει να κάνει όσον αφορά την διαφοροποίηση του ατυχήματος της Φουκουσίμα σε σχέση με το Τσερνομπίλ και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα, τα κατεργασμένα τρόφιμα και κυρίως ε, τα τρόφιμα σε κονσέρβα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Αυτούς τους ομιλητές είχαμε και θα δώσω και πάλι το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνω τις επικρίσεις της κυρίας Ροτμπέρεντ. Θέλω μόνο να διευκρινίσω ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο γιατί δεν είναι η ΕΦΣΑ που μελέτησε. Πρόκειται για τους εμπορεγνώμενες της Ευρατόμ. Και υπήρχε ένα σημείο για τα ψάρια και την πιθανή μόλυνσή τους στον Ειρηνικό ωκεανό. Το συζητήσαμε όταν παρουσιάστηκε αυτό το, το μέτρο στην Ρυθμιστική Επιτροπή και στα κρατημέλη. Έχουμε βάλει μια σύσταση στο σύστημα γρήγορης ενημέρωσης, ε, ε, γρήγορου συνεγερμού, ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να παρακολουθούν και να κάνουν έρευνες ε, σε ορισμένες αλληλευτικές περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους ε, κωδικούς για να ελέγχεται και η είσοδος ε, αυτών των απελευμάτων στην Ένωση. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους αποτέλεσμα για πιθανή μόλυνση των ψαριών σε αυτές τις περιοχές, αλλά τα κράτη-μέλη θα παρακολουθούν από εδώ και μπρος ε, τα ψάρια τα οποία αλλιεύονται σε αυτές τις περιοχές. Τα μέτρα που λάβαμε ε, και υιοθετήθηκαν ε, χθες καλύπτουν και τα ψάρια που αλλιεύονται στην παράκτια περιοχή των περιοχών που καλύπτει ο κανονισμός μας. Τα ψάρια δηλαδή που αλλιεύονται σε αυτές τις περιοχές υπόκειται σε έλεγχο όσον αφορά τη ψάρια δηλαδή τα οποία προορίζονται για εξαγωγή προς την Ευρώπη. Αλλά αυτά είναι τα ψάρια που, που, που αλλιεύονται στις παράκτιες περιοχές. Τώρα, για τα επίπεδα μόλυνσης ε, που περιλαμβάνονται στον κανονισμό 3954. Αυτά είναι κοινά για όλα τα κρατημέλη και γνωστά. Και όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, είναι εμπειρογνώμονες συνθήκες του Ευρατόμ και τώρα του ζητήθηκε να εξετάσουν και πάλι αυτόν τον μέσο όρο και μας υπέβαλαν αυτά τα επίπεδα. Για την ώρα λοιπόν εγώ πρέπει να εργαστώ με αυτά τα επίπεδα ή τον 39-54 είτε αυτό που κάναμε τώρα χρησιμοποιώντας τα επίπεδα τα οποία εφαρμόζονται και στην Ιαπωνία. Τώρα, όσον αφορά τα συσκευασμένα προϊόντα και ιδιαίτερα τα κονσερβοποιημένα προϊόντα, αυτά υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους όπως και οποιοδήποτε άλλο είδος τροφίμου που προέρχεται από την Ιαπωνία από την περιοχή του Ειρηνικού και τις συστάσεις για τα ψάρια, είτε είναι συσκευασμένα είτε είναι κοσυροποιημένα. Εκεί συστήνεται να γίνονται τυχαίοι έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα. Ε, μία σύντομη ερώτηση. Αυτό που ρωτήσαμε και η Τάκμαρ και εγώ είναι ότι δεν μας ικανοποιεί να χρησιμοποιούνται μόνο οι δικοί της Euratom γι' αυτό. Πρέπει να υπάρχουν και ογκολόγοι ή άλλοι γιατροί που ασχολούνται με άλλους τομείς που δεν είναι συνδεδεμένοι με την πυρηνική βιομηχανία. Ποιο ρόλο παίζει η ΕΦΣΑ ή θα παίξει η ΕΦΣΑ και άλλοι εμπειρογνώμονες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με, την με τον πυρηνικό χώρο. Η Κομισιόν. Μιλούσα με τον συνάδελφο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, ο οποίος είναι και ο πιο ειδικό. Αυτοί οι ειδικοί συμπεριλαμβάνουν και τις ειδικότητε που αναφέρατε εσείς. Δεν μιλάμε απλά και μόνο για μηχανικούς, τεχνικούς. Είναι εμπειρογνώμονες που προέρχονται από ένα φάσμα επιστημών. Εμείς ως Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ στην Κομισιόν δεν έχουμε σκοπό να εμπλέξουμε την ΕΦΣΑ σε αυτό. Προς το παρόν. Η Ντάγμαρ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Προηγουμένως μίλησα για την ΕΦΣΑ. Ξέρω ότι δεν είναι ε, αρμόδια, γι' αυτό ε, κοίταζα έτσι με τόσο άγριο βλέμμα προς τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας. Και η ενέργεια ανήκει στην ενέργεια. Το ξέρω. Ε, Εκεί είναι η δυσκολία. Την ΕΦΣΑ την ανέφερα εγώ ως παράδειγμα. Ότι οι επιστήμονες συχνά αντιφάσκουν ή βασίζουν τις αποφάσεις τους και τις γνώμες τους σε στοιχεία αλλά ε, ε, πριν την αρχή της προφύλαξης. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους τους συναδέλφους Επιγόντω και εκείνου τη Γενική Διεύθυνση ενέργεια και τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βεβαιωθούμε ότι ό,τι και αν λένε οι υψηλοί εμπειρογνώμονε τη Ευρατόμ για τι αεροριακέ τιμέ που γίνονται ανεκτέ, πολιτικά δεν πρόκειται ποτέ των ποτών αυτές οι ωραίες τιμές να είναι χαμηλότερες από κάποιες άλλες που να ισχύουν σε άλλες περιφέρειες του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ιαπωνία. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να είναι μια είδηση που να φτάσει παρακαλώ στους αποδέκτες. Διότι άκουσα στο ράδιο Αρβίλα ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξεπλάγησαν ότι δεν θεωρήσαμε σωστή αυτή τη ρύθμιση του Τσερνομπίλ. Γιατί μας ισχύουν λένε οι ωριακές τιμές και τι έγινε, τι πρόβλημα έχετε. Δεν ήταν καν πρόθυμοι να τις χαμηλώσουν ή να ενισχύσουν την ασφάλεια καν. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια είδηση που να φτάσει στους αποδέκτες. Ό,τι και αν μαγειρευτεί εκεί, ποτέ δεν πρόκειται να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που να είναι ε, έστω και κατά διάνοια χαλαρότερο από αυτό που ισχύει στην Ιαπωνία ή αλλού. Ο Βιτόριο Πρόντι. Διευκρίνηση μόνο για ε, το εξής. Γιατί εδώ και κάποιες ε, δεκαετίες ασχολούμαι με αυτά τα θέματα και με την πυρηνική ασφάλεια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής. Και η με ενδιαφέρεται βεβαίως και για την εφαρμογή κάποιων κανόνων. Κανόνων που απορρέουν από φορείς τελείω ανεξάρτητου από τη βιομηχανία. Και αυτή είναι η διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Ραδιενέργεια, που είναι μια επιτροπή τελείω ανεξάρτητη και είχε διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στη διευκρίνηση των μονάδων μέτρησης των ενιών και των κριτηρίων που ισχύουν και που θα πρέπει να ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα δηλαδή και η αρχή της ζημίας ή της βλάβης που προκαλείται, η σωματική βλάβη από τη ραδιενέργεια, αλλά και γενικότερα για πιο χαμηλές δόσεις πρόκειται για ε, πιθανούς κινδύνους, έτσι, είναι κάτι το θεωρητικό στη ζημία του οργανισμού, τη σωματική, δεν έχουμε κάτι, μια βλάβη που να αφορά άμεσα τον οργανισμό εκείνου που έχει εκτεθεί. Ε, και είναι και αναλογική η ε, σοβαρότητα με την έκθεση σε ακτινοβολία. Στα σωρευτικά φαινόμενα η πιθανότητα να ε, αποδειχτεί, μάλλον να προκληθεί ασθένεια είναι αντίστοιχη με την δόση που έχει κανείς απορροφήσει και γι' αυτό ίσως θα πρέπει κάπως διαφορετικά να το σκεφτούμε ακριβώς επειδή πρόκειται για ζημιές οι οποίες άμεσα συνδέονται με την δομή των με τα νουκλεΐδια. Βέβαια αυτές ε, οι έρευνες γίνονται αποκλειστικά ε, προς όφελος μιας επιστημονικής εμπάθεσης και της δυνατότητας ε, αντικειμενικής επιστημονικής άποψης. Έπειτα υπάρχουν διάφορες, διάφοροι οι οποίες, και, και μάλλον τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται για την ε, συνολική προστασία των πληθυσμών και τις οποίες ε, τα οποία μέτρα τα ε, προσπίζει η Ευρατόμα από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομισιόν για τελικέ παρατηρήσεις. Σημειώνω αυτά που είπατε και θα τα διαβιβάσω. Εγώ δεν είμαι ειδικό στην πυρηνική ενέργεια, θα διαβιβάσω το μήνυμά σα. Γνωρίζω απόλυτα αυτά τα οποία είπε η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε σε αυτό το θέμα όταν καταλήγουμε σε επίπεδα ε, διαφορετικά από αυτά που ισχύουν τώρα, αλλά προς το παρόν θα το αφήσουμε στα, στους εμπειρογνώμονες της Euratom. Φυσικά παρακολουθούμε σε τακτική βάση, σχεδόν εβδομαδιαία, τι έλεγχοι γίνονται από τα κράτη-μέλη. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τις Ιαπωνικές αρχές και απευθυνόμαστε και μάλλον ασχολούμαστε και με την ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού σας διαβεβαιώ, από τη στιγμή που θα έχουμε το παραμικρό στοιχείο ότι τα μέτρα που έχουμε είτε δεν λειτουργούν είτε δεν επαρκούν, θα τα επανεξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιστρέψουμε σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, θα τα πούμε το απόγευμα. Γεια σας.